Bene, penso che Μπορούμε να ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας με την ανταλλαγή απόψεων με τον δόκτωρα Κορνέλιο Ζάντεπαρ που είναι μιας ε, Γερμανικού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων μιας γερμανικής εταιρείας που έχει εκπονήσει μια ενδιαφέρουσα μελέτη όχι για όλου. Εν πάση περιπτώσει είναι μια ενδιαφέρουσα μελέτη για το ρόλο και τη σχέση του ειδικού απεσταλμένου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώ είναι υπεύθυνο για αυτό το πεδίο έρευνα που όπω σα είπα συγκεντρώνεται σε αυτό το κείμενο με τίτλο τη εμβάθυνση στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η υπόθεση των, εξωτερικών, των ειδικών απεσταλμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να χαιρετήσω και τον κύριο Ποπόλσκι που θα έρθει από ό,τι κατάλαβα Γενικό Αντιπρόεδρος ε, της ε, υπηρεσίας, ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης θα είναι σύντομα μαζί μας για να συμβάλλει στη συζήτηση. Γνωρίζετε ότι ο ρόλος των ειδικών απεσταλμένων της Ένωσης με την εφαρμογή της Λισαβόνας κάπως αναδιαμορφώθηκε σε σχέση με τις τα καθήκοντα που είχε παλιότερα. Αλλά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης χρειάζεται μια, ένας νέος ορισμός του ρόλου του και αιτιολόγηση του ρόλου αυτού. Και εδώ ακριβώς ε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να το σχολιάσουμε και να δώσουμε υποδείξεις και προτάσεις, ώστε ο ρόλος αυτός να ασκηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ε, ε, λειτουργίας. Δεν έχω τίποτα ακόμα να προσθέσω. Έχετε το λόγο, δόκτωρα Άντεμπεργκ. Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την Επιτροπή ΑΦΕΤ που με κάλεσε να κάνω αυτή την παρουσίαση θα πρέπει να πω πως είναι τιμή μου να σας παρουσιάσω τα απορίσματά μου. Ίσως κάποιοι από σας να γνωρίζετε ότι βασίστηκαν όλα αυτά σε μια διδακτορική διατριβή και πραγματικά ε, αισθάνομαι πολύ ωραία που η έρευνά μου δεν θα μείνει σε έναν χρυσελεφάντινο πύργο. Ε, είναι μεγάλη μου τιμή λοιπόν. Ε, αισθάνομαι πιο περήφανος και πιο ενθουσιασμένος από ότι όταν παρουσίασα τη διατριβή μου την ίδια. σχόλια εκτός μικροφώνου. Ε, θα προσπαθήσω να σας δώσω μια πιο πρακτική προοπτική. Ε, να σας ε, μιλήσω για το θέμα της θέσης μου, δηλαδή το ρόλο του ειδικού εκπροσώπου εντός της Ένωσης. Νομίζω πως ο ρόλο του δικού προστατευόμενου θα πρέπει να οριστεί μέσα στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Σύντομη παρουσίαση, που μου, τα 15 λεπτά δηλαδή που μου δίνονται για να σα παρουσιάσω αυτή την ε, εργασία, θα ακολουθήσω το έγγραφο που σας έχει μοιραστεί, ε, το, όχι το βιβλίο, ε, για το ρόλο των ειδικών απεσταλμένων της Ένωσης και μέχρι στιγμής ε, θα τονίσω την ε, κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, όπου έχουμε από τη μία πλευρά την, εξωτερική, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, ε, που έχει δημιουργηθεί και έχουμε και κάποιες από τις εντολές οι οποίες εκπνέουν στα τέλη του επόμενου μήνα και τέλος θα παρουσιάσω κάποια πιθανά κριτήρια για την επιλογή και τον ορισμό των ειδικών απεσταλμένων και πώς αυτοί μπορούν να εσωματωθούν στην υπηρεσία. Όσον αφορά το πρώτο μου παρατήρηση, το ιστορικό ε, αυτοί έχουν αποκληθεί ως ε, το πρόσωπο της Ένωσης στο εξωτερικό, έχουν ασχοληθεί με την επίλυση κρίσεων σε διάφορα περιοχές ενδιαφέροντος για την Ένωση. Στην πράξη δηλαδή έχουν βοηθήσει στη διευκόλυνση ειρηνευτικών συνομιλιών, έχουν επιβλέψει συμφωνίες ανάμεσα σε εμπόλεμα μέρη, έχουν ε, προωθήσει διεθνείς διαπραγματεύσεις μαζί με άλλους εταίρους και έχουν δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 15 χρόνια πληροφορίες από τι συγκεκριμένε περιοχέ, πληροφορίε που διαφορετικά δεν θα είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δύο ειδικοί, οι πρώτοι ειδικοί εκπρόσωποι είχαν στην αποσταλή το 1996 και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 11 εντολέ σε διάφορε περιοχέ ε, ε, του κόσμου. Τώρα, η ετολόγηση ε, υπάρχει ένα ευρύ πλαίσιο το οποίο βασικά σχετιζόταν με την ιδέα του να δοθεί πολιτικό βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μέχρι τότε είχε περισσότερο οικονομικό βάρος σε ορισμένε περιοχές να δίνει πληροφορίες για μια συνεχιζόμενη σύγκρουση επιτόπου και να, να ξεκινά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, η διαμεσολάβηση και να δίνει πολιτικές συμβουλές. Ε, εκτός από αυτή την ε, λειτουργία η οποία ήταν στραμμένη προς το εξωτερικό είχε και μια σημαντικό ρόλο στο να γεφυρώνει ε, τις, τα κενά ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές ανάμεσα δηλαδή στην ΚΕΠΑ την Ένωση αλλά και τις επιτόπου αποστολές των ειδικών απεσταλμένων αλλά και, ανάμεσα στον, και, με τον δεύτερο πυλώνα γιατί συνεργάζονταν με την Ευρωπαϊκή Κομισιόν σε πολλές πολιτικές ε, όπως ε, στην γυρνίαση ή στην πρόληψη συγκρούσεων. Αυτά λοιπόν για να σας πω ότι ένας απεσταλμένος είναι μια, ε, ένα φυσιολογικό διπλωματικό εργαλείο χρησιμοποιείται από άλλους οργανισμούς όπως ο ΙΕ, άλλα κράτη σε ολόκληρο τον κόσμο η ΙΠΑ. είναι μια τέτοια περίπτωση που εξέτασα αλλά και από τα ίδια τα κράτη-μέλη ακόμα και στις περιοχές όπου ήδη υπάρχουν ειδικοί απεσταλμένοι της Ένωσης. Ορισμένοι θεωρούν πως είναι ένα απαραίτητο μέσο για επιτυχή διπλωματίας στη σημερινή περίπλοκη κατάσταση. Αυτή ήταν η πρώτη λοιπόν παρατήρηση όσον αφορά την εξέλιξη των 15 χρόνων ύπαρξης των ειδικών απεσταλμένων και της ευρωπαϊκής σχετικής πολιτικής. Τώρα, ε, δεύτερη μου παρατήρηση είναι ότι υπήρξε μια μεγάλη αλλαγή που προέρχεται από, ρέη από την συνθήκη της Λισαβόνας και συνδέεται άμεσα με τους ειδικού απεσταλμένους. Ε, σύμφωνα με την προηγούμενη εκδοχή της συνθήκης, εκεί έλεγε ότι το Συμβούλιο μπορεί να ορίζει έναν ειδικό απεσταλμένο όποτε το θεωρεί απαραίτητο. Δηλαδή εξαρτάται από το Συμβούλιο, από τα κράτη-μέλη που έθελαν να στείλουν έναν ειδικό απεσταλμένο ή αν δεν ήθελαν. Το νέο άρθρο 33 της Συνθήκης της Λισαβόνας λέει ότι το Συμβούλιο μπορεί να ορίσει έναν ειδικό απεσταλμένο μετά από πρόταση του είπα το εκπροσώπου. Μεγάλη αλλαγή αυτή γιατί το Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ειδικό απεσταλμένο μόνο αν ο, ειδικό, ο είπατος εκπρόσωπος το προτείνει. Οπότε αυτό είναι κάτι που ήταν κρίσιμο σημείο και για την Ε, σημερινή κατάσταση που όπως σας είπα εκπνέουν κάποιες εντολές τον επόμενο μήνα. Το... Αυτό που θα συμβεί είναι ότι ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θα αναλάβει κάποιε από τι ε, λειτουργίε που είχαν οι ειδικοί απεσταλμένοι μέχρι στιγμή. Γι' αυτό και στι σημερινέ εντολέ υπάρχει κάτι το οποίο ονομάζεται ε, sunset clause, δηλαδή είχαν συγκεκριμένη ημερομηνία τέλο, αλλά θα μπορούσαν και να κλείσουν νωρίτερα οι εντολέ αν η λειτουργία ε, αυτών των ειδικών απεσταλμένων, ο ρόλος τους μπορούσε να αναλυφθεί από την εξωτερική υπηρεσία. Ε, τώρα, Είπατε εκπρόσωπος και τα κράτη-μέλη που αντιπροσωπεύονται στην Πολιτική Επιτροπή και στην Πολιτική Ασφάλεια ξεκίνησαν πριν από ένα χρόνο Συνήθως οι εντολές ε, διαρκούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, οπότε πριν από ένα χρόνο ξεκίνησε η συζήτηση ανάμεσα στον ΙΠΑ, το εκπρόσωπο και την ε, εξωτερική υπηρεσία για να δουν ποιες ε, εντολές θα πρέπει να συνεχιστούν. Υπήρξε μια πρώτη κλιμάκωση το περασμένο καλοκαίρι και εξευρέθη μια συμβαστική λύση ανάμεσα στην ΕΠΑ το εκπρόσωπο ήθελε να κλείσει κάποιες από τις εντολές και τα κράτη-μέλη που δεν το ήθελαν αυτό τότε. Ευρέθη λοιπόν μια συμβαστική λύση ώστε τέσσερις εντολές να επεκταθούν ε, για ακόμα μισό χρόνο μέχρι το Φεβρουάριο δηλαδή, και ορισμένε άλλε εντολές ε, ε, παρατάθηκαν μέχρι τον Αύγουστο του τρέχοντος ε, έτους. Έχουμε δηλαδή Μολδαβία, ειρνευτική διαδικασία Μέση Ανατολή, Νότιο Κάφκασο και Κωσυφοπαίδιο που θα κλείσουν τώρα το Φεβρουάριο, εκτό και αν παραταθεί η εντολή του. Εκτό δηλαδή και αν είπα του εκπρόσωπου σου προτείνει να παραταθούν οι εντολέ. Γιατί όπω είπα, το Συμβούλιο το ίδιο δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Το ερώτημα είναι τώρα λοιπόν, αυτές οι τέσσερις εντολές είναι αυτές που θα μπορούσε να αναλάβει η ίδια η εξωτερική υπηρεσία. Άμεσα. Έχουν σχέση με, δηλαδή τις χρειαζ, ξεκολουθούμε να χρειαζόμαστε αυτές τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Και έπειτα, ποια είναι τα πιθανά κριτήρια για το πότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσει δικούς απεσταλμένους η Ένωση και αν το αποφασίσει πώς θα πρέπει αυτοί να συνεργάζονται με την εξωτερική υπηρεσία και αν τελικά αποφασιστεί να τελειώσει μια εντολή ενός απεσταλμένου πώς θα λειτουργήσει και πώς θα διαχειριστούμε την μεταβατική περίοδο γιατί αυτό που έχει καταστεί σαφές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι ότι δεν είναι μόνο τεχνικό το θέμα, δεν είναι απλώ να πούμε εντάξει τελειώνει μια εντολή, ούτως ή άλλω είχε ημερομηνία λήξη και θα λήξει αυτομάτως. Ιδιαίτερα οι πιο μακροχρόνιε εντολέ και οι 11 εντολέ των ειδικών απεσταλμένων ισχύουν εδώ και χρόνια Πράγμα το οποίο δημιουργεί προσδοκίες εξ ονόματος των διεθνών εταίρων, από πλευρά των διεθνών εταίρων οργανισμών, αλλά και των κρατών που έχουν τους ίδιους ε, τους, τους ειδικούς απεσταλμένους, όπου γίνονται διαπραγματεύσεις κτλ. Αυτό δημιουργεί προσδοκίες σε σχέση με την δέσμευση της Ένωσης επιτόπου, με τα Ε, κράτη-μέλη δημιουργούνται, προκαλούνται αρνητικές αντιδράσεις των ίδιων των περιοχών, εκεί όπου αμφισβητείται δηλαδή η εντολή κάθε φορά το ειδικό απεσταλμένο. Τώρα όσον αφορά τα κριτήρια και αυτό που θα, θέλ, θέλω να σας παραπέμψω και στο φυλάδιο που σας έδωσε. Υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος, σχετικά μακρύς κατάλογος για τα κριτήρια που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη στρατηγική χρήση των απεσταλμένων. Όταν υπάρχουν ήδη διεθνείς ε, οργανισμοί που ασχολούνται για την επίλυση κρίσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη περιοχή και δεν θέλει να βρίσκεται εκεί μόνο για βράχη πρόθεσμα, ε, Τώρα, το είδος του προσωπικού που επιλέγεται για να λειτουργήσει ως ε, ειδικό απεσταλμένο ε, θα πρέπει επίσης να εξεταστεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας κατάλογος που δεν ε, είναι η βίβλο, αλλά που θα πρέπει να μας αποτελέσει μια βάση για την συζήτηση. Ώστε η συζήτηση αυτή να γίνει σε σχέση με τους στόχους που θέλει να πετύχει η Ένωση σε κάθε τέτοια περιοχή. Ε, αν αρκεί δηλαδή αυτό το, το μέσο το ειδικό, του ειδικού απεσταλμένου ή όχι. Το θέμα προκύπτει αν χρησιμοποιήσουμε ε, τα κριτήρια αυτά και εξετάσουμε τις σημερινές εντολές, κάποιες από τις σημερινές εντολές ε, θα μπορούσαν να εκλείψουν. και αυτό σχετίζεται με το πώς η Ένωση θα οργανώσει την μεταβατική περίοδο. Και αυτό είναι κάτι που, όπως σας είπα, η Ένωση θα πρέπει να δει όχι ad hoc, αλλά σε στενή συνεργασία με τα, τις ενδιαφερόμενες χώρες και τις χώρες εταίρους. Μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου πιθανότατα όμως δεν θα προλάβει να το κάνει. Δεν γίνεται να υπάρξει ένα phase out των ισχυούσων εντολών. Και έπειτα, αν συνεχιστούν οι εντολέ, και εγώ πιστεύω πω πολλέ από αυτέ θα πρέπει να συνεχιστούν, πώ αυτέ θα ενταχθούν στην εξωτερική υπηρεσία. Εδώ υποβάλλω κάποιε προτάσει σε σχέση με την δομή στήριξη. Αυτή τη στιγμή οι 11 οι ειδικοί απεσταλμένοι έχουν τη δική τους υποστήριξη, δηλαδή διοικητική, λογιστήρια κτλ. Αυτά εύκολα μπορούν να ενσωματωθούν στην εξωτερική υπηρεσία. Το θέμα των πολιτικών συμβούλων προκύπτει. Αν δηλαδή οι σημερινοί μπορούν να μεταφερθούν στην εξωτερική υπηρεσία ή αν οι μελλοντικοί πολιτικοί σύμβουλοι θα πρέπει να αντληθούν από την εξωτερική υπηρεσία. Εν πάση περιπτώσει όμως τελικά το ε, μέσο του ειδικού απεσταλμένου είναι σκόπιμο, κέριο και πρόκειται για ένα μέσο το οποίο βασίζεται σε ένα άρθρο της συνθήκης και πιθανότατα είναι, και είναι κάτι το οποίο άμεσα συνδέεται με τον ύπατο εκπρόσωπο και ίσως, όπως βλέπετε και από το οργανόγραμμα, είναι έξω από την δομή της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Υπηρεσίας. Για να ολοκληρώσω, όπως σας είπα, ο ειδικό επεσταλμένος είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο στη διπλωματία και στην επίλυση συγκρούσεων τη σήμερων ημέρα. Είναι κάτι που έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του τα τελευταία 15 χρόνια και πιστεύω, και επανέρχομαι στα όσα είπα στην αρχή, ότι το διδακτορικό μου σχετιζόταν με αυτό το θέμα ήταν ε, ένα δεκτορικό για πολιτικές επιστήμες, αλλά πολλοί με πλησίασαν και μου είπαν ε, γιατί να μην γράψεις ε, δεκτορικό ιστορικό αφού σύντομα θα καταργηθούν οι δικοί επισταλμένοι. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι τέτοιο και προσβλέπω στη συζήτηση μαζί σας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Μπράτνερ. Εγώ θα μιλήσω γερμανικά. Τρελώνει το να μιλάμε με Γερμανοί μεταξύ μας αγγλικά. Ε, χάρηκα πάρα πολύ που ε, βρήκα το χρόνο να έρθετε εδώ και να παρουσιάσετε τη μελέτη σας. Ε, βεβαίως ε, είχαμε διαβάσει προηγουμένως τα στοιχεία που σας αφορούν. θέλω όμως να πω, υπάρχουν κάποια δύσκολα θέματα αυτή την εποχή. Το Κοσφοπέδιο, η Βοσνία. Μήπως μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα πώς βλέπετε την ε, κατάσταση ε, στο κοσυφοπέδιο ε, μήπως θα πρέπει να παραταθεί η παραμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην επέλθει το χάος όμως και το θέμα της στρατηγικής που δεν έχει διευκρινιστεί. Ποια είναι η δική σας η άποψη από αυτού. Και κάτι άλλο, ίσως ένα σχόλιο που αφορά στην εργασία σας, δηλαδή ποιες γνώσεις θα πρέπει να έχει ένας ειδικό απεσταλμένος. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει και ικανότητες στη διαχείριση των κρίσεων και στις ε, διαπραγματεύσεις. Ε, είναι σημαντικό αυτό, γιατί αν ε, περιγράφει κανείς τα καθήκοντα, όπως το κάνετε, κάτω από το πρίσμα της επεξεργασίας των περιφερειακών συγκρούσεων, των διασυνοριακών πάλι συγκρούσεων. Ε, τώρα όμως ε, είναι σημαντικότερο να έχει κανείς και άλλες ικανότητες. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με αυτό που είπατε. Πράγματι θα τους χρειαστούμε τους ειδικού απεσταλμένους ε, και στο μέλλον. Και τίθεται το εξής ερώτημα αυτός ο special envoy, όπως τον λέμε στα αγγλικά, Χρειάζεται πράγματι, δηλαδή να έχει βραχυπρόθεσμα, να λαμβάνει κάποια εντολή. Να πηγαίνει, ας πούμε, τώρα στην Τινησία ως ε, special envoy ε, και να έρχεται σε επαφή με την κοινωνία. Όχι δηλαδή ε, ειδικό ε, εκπρόσωπος που μένει πολύ χρόνο, να είναι εντεταλμένος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τι είδους δυνατότητες υπάρχουν λοιπόν έτσι ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε ε, σε επίκαιρα θέματα. Πάντως όσον αφορά τη γενικότερη ανάλυση σας συμφωνώ απόλυτα. Ευχαριστούμε. Μούνιτς. Κυρία Μούνιτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εμένα με εντυπωσιάζει κάπως ε, η ένταση με την οποία υπερασπίζεστε την... Ε, τις επικρίσεις ε, τις οποίες υποβάλλατε έναντι της είπα της εκπροσώπους. Είπα της εκπροσώπου για τη δυνατότητα δηλαδή να μην ανανεωθούν, την πιθανότητα να μην ανανεωθούν εντολές διαφόρων ειδικών απεσταλμένων. Εγώ πιστεύω ότι έχουν παίξει χρήσιμο ρόλο όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε άλλους, ε, άλλα μέσα στη διάθεσή της ε, όπως έχει τώρα δηλαδή την εξωτερική υπηρεσία. Νομίζω πως οι ειδικοί επεσταλμένοι είναι προβλέπονται στη συνθήκη, αλλά στην ουσία είναι μια υπενθύμηση του αδιέξοδο της διακυβερνητικής ε, αυτής κατάστασης που στόχο έχει να γίνει κοινοτική πολιτική. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει στο μέγιστο δυνατό βαθμό να χρησιμοποιείται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης, ε, να ενισχυθεί και να ε, επανδρωθεί με τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους και τους πολιτικούς πόρους, ώστε να ολοκληρώσουν, να κλείσει πια αυτή η υπόθεση των ειδικών απεσταλμένων. Κατά δεύτερο λόγο θα ήθελα ε, μάλλον εσείς είπατε ότι η ανάγκη ύπαρξης ε, ειδικών απεσταλμένων ε, συνήθως ε, παληθεύεται σε περιπτώσεις ε, σύγκρουσης. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνεται αυτό με οριζόντιο χαρακτήρα, όχι μόνο για περιπτώσεις ε, σύγκρουσης, ε, για θέματα όπου η Ένωση τα αντιμετωπίζει με άλλα μέσα, όπως το μέσο της σταθερότητας, θα μπορούσαν πούμε, να χρησιμοποιηθούν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στα θέματα οικοδόμησης της ειρήνης, με στόχο στοχοθέτηση πιο προσανατολισμένη στη συνεργασία. Θα πρέπει λοιπόν να Θα πρέπει λοιπόν η εξωτερική υπηρεσία που θα είναι η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να συγκρίνεται με τη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ. Εμείς ε, προσβλέπουμε να παίξουμε πλήρη ρόλο στη διεθνή σκηνή και όχι να είμαστε μια γενική υπηρεσία που να θέλει να λύσει κάποιες συγκεκριμένες συγκρούσεις. Ευχαριστώ. Κυρία Λούζινγκ, ευχαριστώ πολύ. Ε, Αντεμπά, ε, το βιογραφικό σας αναφέρεται και το είπατε κιόλας ότι τώρα πλέον η αρμοδιότητα για τους ειδικού απεσταλμένους ε, είναι στα χέρια της κυρίας Άστον. Και δεν είμαι σίγουρη για, τι σημαίνει, για το τι σημαίνει αυτό, αλλά θέλω να σας ρωτήσω μήπως ε, αυτό θα οδηγούσε στο να διαμορφωθεί διαφορετικά ο κοινοβουλευτικό έλεγχο πάνω στου ειδικού απεσταλμένου. Επ' αυτού θα ήθελα να έχω τη γνώμη σα. Ε, και κάτι άλλο για την στρατηγική ε, συγκρούσεων και σειράξεων. Ε, προτάθηκε οι ειδικοί επεσταλμένοι ε, στο μέλλον ε, να έχουν επίκαιρα ε, προγράμματα έκτακτης ανάγκης. Κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ένα παράρτημα όπου να αναφέρεται και το ενδεχόμενο της στρατιωτικής επέμβασης. Εσείς λοιπόν αυτή την πρόταση πώς την κρίνετε και πιστεύετε ότι στις μελέτες σας για την στρατηγική ε, συγκρούσεων μπορεί να συμπεριληφθεί και αυτό το θέμα της ε, στρατιωτικής επέμβασης. Λαντστοφ, επόμενη ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να φερθώ σε ορισμένα που ελέγχθησαν από τους συναδέλφους και να υπογραμμίσω ότι κατά τη δική μου άποψη αυτό το εργαλείο του ειδικού απεσταλμένου σε επίπεδο αρχής είναι ένα καλό εργαλείο, μια καλή δυνατότητα. Όμως τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Εγώ το βλέπω διαφορετικά από ό,τι το έθιξε η κυρία Μούνιτς. Δηλαδή το ερώτημα που τίθε δεν είναι αν θα υπάρχει ειδικό απεσταλμένος ή υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Το πρόβλημα που έχουμε με την κυρία Άστον είναι ότι έχουμε μία ύπατη εκπρόσωπο η οποία ακριβώς ε, όπως και άλλοι Υπουργοί Εξωτερικών δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα του να είναι πανταχού παρόντες. Δεν μπορεί να είναι πανταχού παρούσα. Χρειάζεται λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χρειάζεται και μία εκπροσώπηση σε πολιτικό επίπεδο σε περιοχές κρίσεων, προφανώς για οριζόντια θέματα, δεν ε, το αμφισβήτω αυτό. Δείτε λοιπόν το εξής ερώτημα. Μήπως στο μέλλον τέτοιου είδους ε, ειδικοί απεσταλμένοι πρέπει να είναι πολιτικοί εκπρόσωποι όπως συνέβη, ας πούμε, συμβαίνει στην Αμερική, ο κ. Μίτσελ, οι γερουσιαστές. Να είναι λοιπόν πολιτική σύμβουλη. Αυτό είναι πολύ πιο λογικό από το να συνεχίσουμε με τους επαγγελματίες καριέρας. Γιατί αυτοί υπάρχουν οι επαγγελματίες καριέρας, εντάσσονται στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και δημιουργούνται προβλήματα τριβής με αυτούς. Τώρα, πάω σε ένα άλλο θέμα που συμφωνώ με την Μαρία Μούνιθ. Πράγματι, το Συμβούλιο μετά από εκπρόσωπο, με συγχωρείτε, μετά από συμβουλή ε, σύσταση της ύπαρξη εκπροσώπου ορίζει έναν ειδικό αντιταλμένο, ο οποίος όμως λειτουργεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο του Συμβουλίου. Βέβαια, αυτή η διαδικασία ε, πρέπει να περάσει από το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό είναι απαραίτητο. και θα μπορούσε ίσως ε, η ύπατη εκπρόσωπος να ορίζει και δικούς της απεσταλμένους γιατί αυτή έχει ε, και άλλους πόρους ε, στη διάθεσή της. Υπάρχει λοιπόν το εξή θέμα. Οι απεσταλμένοι αυτοί να είναι πιο πολιτικά πρόσωπα, να είναι πολιτικοί σύμβουλοι και να μπορεί η κυρία Άστον να τους διορίζει. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η βελτιστοποίηση της ένταξης μέσα στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης πρέπει ακόμα ε, να επιτευχθεί. Δεν έχει επιτευχθεί. Εν τω μεταξύ, ευχαριστούμε πολύ. Έχει έρθει ο αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα ε, της Υπηρεσία εξωτερικής δράσης, ο κύριο ε, Ποπόφσκι. Γι' αυτό λοιπόν δεν ξέρω τώρα, να παρέμετε και εσείς στη συζήτηση ή να περιμένουμε να ακούσουμε την απάντηση του κυρίου Αντεμπάρ. Εσείς δεν ακούσατε τη δική του την εισαγωγή, γι' αυτό να αποφασίσετε μόνο σας. Θέλετε να μιλήσετε τώρα ή να μιλήσετε μετά, αφού θα έχετε ακούσει τι απαντήσει του κύριου Αντεμπαρ. Τι θέλετε να κάνετε, παρακαλώ, σα ερωτώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, επειδή έχω διαβάσει το έγγραφο, μπορώ να μιλήσω τώρα. Ε, έχω δηλαδή ενημερωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου αποστήλετε. Είναι πολύ έγκαιρη συζήτηση. Ξεκινώντας να πω ότι δεν είναι τόσο αρνητικά τα πράγματα όπως φαίνονται. Οι συζητήσεις συνεχίζονται, συζητάμε τώρα αυτό το λεπτό θέμα με τα κρατη αλλά θα ήθελα να φτάσουμε στην καλύτερη το δυνατόν συστημική λύση τώρα. Κάνοντας το ιστορικό θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι πρόκειται στην ουσία για έναν παλαιό δεύτερο πυλώνα. Η εντολή ε, περιορίζεται στα θέματα ΚΕΠΑ και σε ζητήματα που άπτονται της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας και μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο μέλλον. Θα επανέλθω όμως. Κάτι άστον πιστεύει ότι επειδή έχουμε τη νέα υπηρεσία μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε για διάφορα καθήκοντα τα οποία μέχρι τώρα είχαν λάβει οι ειδικοί απεσταλμένοι. Και έχουμε δύο δυνατότητες. Έχουμε ε, κάποιον ε, επικεφαλής αντιπροσωπείας που θα φέρει φοράει δύο καπέλα. Ε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος έχει τρία καπέλα Καμπούλ, ε, ε, Σκόπια και Αντισαβέμπα. Λοιπόν, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί κατά πόσο θέλουμε να διαδραματίσει έναν εξειδικευμένο ρόλο ή όχι. Όπως συμβαίνει με το θέμα της ειρήνευσης στην Μέση Ανατολή και των ειδικό απεσταλμένο μας. Όπως γνωρίζετε, έχουν μια σειρά από διοικητικούς διευθυντές που έχουν περιφερειακές και θεματικές ε, αρμοδιότητες, αλλά μπορούν επίσης να αναλάβουν και κάποια καθήκοντα που τους ανατίθενται από την είπατε Και ίσως τους προσεχείς εβδομάδες ή μήνες ε, τα κάποιες εντολές θα εκπνεύσουν όπως αυτή που αφορά τον Νότιο Κάφκος και την Μολδαβία. Αναφέρθηκα στον δεύτερο πυλώνα ως βάση για τους ειδικούς απεσταλμένους επειδή η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, έχει έναν ευρύτερο σκοπό, στόχο. Φυσικά είμαστε ένα generis όργανο, το γνωρίζετε καλά αυτό, έγιναν διαπραγματεύσει ανάμεσα στην Καθηνά και το Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά έχουμε και αυτή την ιδιαίτερη, ιδιαίτερο σύνδεσμο με την Κομισιόν. Όταν ε, λοιπόν οι ειδικοί απεσταλμένοι ε, αναλαμβάνουν καθήκοντα, είναι πολύ στενά συνδεδεμένοι με την Κομισιόν αυτή Συμφωνούμε λοιπόν ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ε, υπηρεσία μας και η όλη δομή θα πρέπει να υπάρχει εντός της υπηρεσίας. Αυτό και έχει κάποιες επιπτώσεις δημοσιονομικές που ενδιαφέρουν και το Κοινοβούλιο για τις δραστηριότητες ε, των ειδικών πιστευμένων μέχρι τώρα πλούν από τον προβλησμό της ΚΕΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι δαπανούσαμε σημαντικά ποσά για το προσωπικό και τώρα θα προέρχεται από ένα διαφορετικό, μια διαφορετική θέση στον προπολογισμό. Αλλά θα φροντίσουμε να το ρυθμίσουμε Φυσικά πρέπει να επιλύσουμε τα άμεσα προβλήματα, κάποιες ε, εντολές που θα εκπνεύσουν στο τέλος ε, ε, του έτους. Ε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις επόμενες εντολές, τους ψυχούς μήνες, ή εβδομάδες, σε περίπτωση που εκπνέουν τον θέρος. Αλλά δεν βρισκόμαστε στο τέλος του δρόμου. Υπάρχουν οι περιφερειακές εντολές, πρέπει να αποφασίσουμε το ζήτημα των ειδικών απεσταλμένων, του ειδικού απεσταλμένου για την περιοχή των μεγάλων λιμνών. Και επίση πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα ο ειδικό απεσταλμένος στην Πρετόρια. Δεν αποκλείω νέε ε, εντολές να δοθούν σε ειδικού απεσταλμένου, Συζητείται π.χ έχουμε κάποιον ειδικό απεσταλμένο για το κέρας της Αφρικής. Και αυτό λόγω της δέσμευσης που έχουμε λάβει στην περιοχή, αλλά και για την επιχείρηση Αταλάντη. Τώρα πώς θα πρέπει να διορίζονται οι ειδικοί επισταλμένοι, αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Πρέπει να φροντίσουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ ότι η μορφή έχει ιδιαίτερη σημασία. Όταν υπάρχουν συζητήσεις λοιπόν στην Μέση Ανατολή πρέπει να είμαστε παρόντες. Προεβδομάδος ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής ε, της ε, υπηρεσίας μας ε, εκπροσώπησε την καθιάστον εκεί. Δεν προσπαθώ να βρω μια λύση, αλλά σας λέω ότι είμαστε παρόντες, δεν παραμαλούμε την δυνατότητα να εμπλεκόμεθα σε υφιστάμενες ε, οργανώσεις ε, Φυσικά στο πλαίσιο των περιορισμένων πόρων που έχουμε στην ε, διάθεσή μας Οι ε, περιφερειακές εντολές ε, είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε και θα επανέλθουμε. Φυσικά χρειάζεται να εξετάσουμε και το ζήτημα της ε, συμμετοχής του ειδικού απεσταλμένου στο πλαίσιο της επιχειρήσεων που γίνονται σε περιοχές ε, αρμοδιότητας, π.χ. Καμπούλ, όπου ο ειδικό απεσταλμένο μας ε, συνεργάζεται στενά με την αποστολή της UPOL ε, για την εκπαίδευση της αστυνομίας. Φυσικά πρέπει να επιλύσουμε και τα τρέχοντα προβλήματα, όπως αυτό της εκπνοής των εντολών. Οι συζητήσεις συνεχίζονται αλλά είπα ότι ο πρόσωπος ε, θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο που παρέχει η συνθήκη για να βελτιώσουμε τις ε, σχέσεις ε, μεταξύ της υπηρεσίας μας αλλά και των διαφόρων αποστολών μας που υπάρχουν. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, τα τελικά σχόλια βεβαίως ε, ανήκουν στον εμπειρογνώμονά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, ε, για τις αντιδράσεις σας και ευχαριστώ επίσης και για την παρουσίαση του κυρίου Ποπόφσκη. για μένα είναι μεγάλη τιμή το να μπορώ να βρίσκομαι σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτό το επίπεδο. Θα ήθελα τις απαντήσεις μου να τις ε, στοχεύσω. Καταρχήν ε, την ερώτηση ε, τι είναι ο ειδικό απεσταλμένο και τι είναι οι προσωπικοί απεσταλμένοι, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τα θέματα. Το ευρύτερο θέμα, ποια είναι η στρατηγική που μπορεί να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια συγκεκριμένη περιοχή κρίσης. και τέλος, ο ενδυνάμει ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως είπατε και ορισμένοι από εσά, οι ειδικοί επισταλμένη είναι εργαλείο ε, της συνθήκης και της ΚΕΠΑ. Πράγματι υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό. Αλλά εφόσον θα συνεχίσει να υπάρχει η ΚΕΠΑ, ε, υπάρχει και κάθε λόγος οι ειδικοί απεσταλμένοι να συνεχίσουν να υπάρχουν ακόμα και αν είναι ο δεύτερος πυλώνας όπως το χαρακτήρισε Συμφωνώ με τον κύριο Λάμπστροφ ότι οι δύο θα πρέπει να μπορούν να υφίστανται παράλληλα. Αυτά όταν μιλάμε για έναν ειδικό απεσταλμένο ως ένα επίσημο εργαλείο. Όταν μιλάμε για ε, απεσταλμένους για σύντομο χρονικό διάστημα, για ένα συγκεκριμένο θέμα, ούτε καν για κρίση, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Και μέχρι τώρα έτσι ήταν τα πράγματα. Ο κύριος Σολάνα είχε κάποιους προσωπικούς απεσταλμένους του, οι οποίοι ήταν μέλη ε, του ε, γραφείου του και είχαν έτσι ένα ειδικό τίτλο. Η ύπατη εκπρόσωπος προφανώς είναι ελεύθερη να ορίζει ε, προσωπικό από την υπηρεσία της για τέτοιου είδους θέματα. Εάν όμως επιθυμούμε ένας επίσημος απεσταλμένος να αναλαμβάνει και κάποια θέματα, εκεί θα πρέπει να υπάρχει σαφή οριοθέτηση των αρμοδίτων. Δεν μπορεί να υπάρχει δικό απεσταλμένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ίσω να υπάρχει ένα για τη μη διάδοση των όπλων, αλλά και αυτό οριακά. Ε, η δουλειά, οι αρμοδιότητε των ειδικών απεσταλμένων θα παραμένουν μέσα στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ και της διαχείρισης κρίσεων. Να είναι πολιτικά πρόσωπα, ναι. Αυτό συζητιέται εδώ και πολύ καιρό. Και περιέργως πως στην αρχή είχαμε, στην αρχή δηλαδή της δεκαετίας του 90, είχαμε ε, περισσότερους ε, πολιτικούς ε, απεσταλμένους. Αυτό βέβαια δημιουργούσε δυσκολίες και έτσι προτιμήθηκε να επιλέγονται πάλι της Ευρωπαϊκή Ένωσης οι πρέσβεις, γιατί αυτοί δεν έχουν τόσο, δεν επιμένουν τόσο στις απόψεις τους, ε, κάμπτονται πιο εύκολα. Αυτό βέβαια δεν είναι προσβολή, ε, δεν θέλω, που δεν είναι να προσβάλλω κανέναν. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν τώρα έχουμε διπλωμάτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών που λειτουργούν παράλληλα. Εγώ λοιπόν μπορώ να προβλέψω ε, μια εξέλιξη όπου οι ειδικοί επιστελμένοι αποκτούν περισσότερες πολιτικές αρμοδιότητες και πάλι, για τους λόγους που ανέφερα. Τα τελευταία μας χρόνια σας είπα η τάση ήταν αντίστροφη. Δηλαδή αυτοί ε, εντάχθηκαν περισσότερο στο ε, διπλωματικό σύστημα το ερώτημα των ειδικών απεσταλμένων με δύο ιδιότητες ε, πράγματι ε, αυτή είναι η πρώτη επιλογή αλλά όπως είπε και ο κύριος Μπραντνα ε, στη Βοσνία Ρισεγοβίνη και στο Κωσυφοπέδιο τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά εκεί είναι χώρες όπου οι ειδικοί επεσταλμένοι μπορούν να αποκτήσουν διπλή ιδιότητα. Αλλά υπάρχουν άλλε περιπτώσει που δεν ισχύει αυτό. Και οι λόγοι έχουν να κάνουν με τη δομή της χώρας δομή της ε, συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοια που και κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει κάθε λόγος να συνεχίσουν αυτές οι αρμοδιότητες. Παράλληλα όμως ε, να εξετάζεται και το θέμα των ε, διπλών αρμοδιοτήτων. Το ευρύτερο θέμα της στρατηγικής αντιμετώπισης κρίσεων εγώ δεν εννοούσα ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι ε, θα πρέπει να δουλεύουν με έκτακτα προγράμματα για στρατιωτικές επεμβάσεις. Όχι. Ήδη έχουμε 11 εντολές Άρα δηλαδή θα πρέπει να οριστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτοί, ποιοι είναι οι στόχοι ε, που ε, διεκδικεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες είναι οι σχέσεις ε, με τους ειδικούς απεσταλμένους. Το να ζητάμε να υπάρχει ένα τέτοιο έγγραφο που να περιλαμβάνει στοιχεία πρόληψης κρίσεων, το να ζητάμε να υπάρχει ένα τέτοιο έγγραφο ε, οποτεδήποτε ορίζεται και ένας νέος απεσταλμένος, αυτό γιατί όχι. Αυτό έχει σχέση και με το ερώτημα που τίθεται επιτάπητος, δηλαδή εντολές ε, που θα εκπνεύσουν ε, τον επόμενο μήνα. Ομολογώ ότι προσπαθώ να πιστώ γιατί πρέπει να εκπνεύσουν αυτές οι εντολές. Δύο, στην αρχή ήταν τέσσερις μάλιστα. Φαίνεται ότι εκεί έγινε μια επιλογή. Και γι' αυτό το λόγο προσπάθησα να βρω κάποια κριτήρια. Μια λογική. Βεβαίως και υπάρχει λόγος να εκπνεύσουν κάποιες εντολές. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνεται και με κάποια λογική. Και όχι έτσι παρορμητικά ή ad hoc, γιατί ήδη διαφαίνονται κάποιες επιπτώσεις. Και τέλος, Τώρα, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πράγματι ε, έχει τη δυνατότητα ε, εδώ να ανταλλάσσει απόψει ε, και να ανταλλάσσει απόψει το Κοινοβούλιο με του ειδικού απεσταλμένου πριν αυτοί να λάβουν τι αρμοδιότητέ του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί βέβαια να καλέσει όλου του ειδικού απεσταλμένου να έρθουν εδώ και να μιλήσουν. Πάντω αυτό που ισχύει για το Κοινοβούλιο που έχει λόγο για τους επικεφαλεί αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει λόγο το Κοινοβούλιο και για του ειδικού απεσταλμένου. Υπάρχει λοιπόν ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η κυρία Άστον όπως ξέρετε λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο Αυτά ε, νομίζω είναι αυτά που είχα να σα πω. Θα παρακολουθήσουμε πολύ ενδιαφέρον το πώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει το ρόλο του και πώ το εργαλείο αυτό των ειδικών απεσταλμένων, το Κοινοβούλιο ε, θα το ε, εντάξει περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρότι με βάση τη συνθήκη παραμένει ένα διακυβερνητικό εργαλείο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντεμπάρ. Υπάρχει κάτι ακόμα που θέλει να πει όμως ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγγνώμη έχασα την αρχή της συζήτησης. Είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει ρόλος ε, για τους ειδικούς απεσταλμένους να συντονίζουν τις εργασίες σε περιφερειακό επίπεδο και να ξεπερνούν ε, τα ε, εδαφική επικράτεια του κράτους το οποίο είναι εγκαριστημένοι. Υπάρχει και ρόλος φυσικά και για βουλευτές και για κάποιους ακαδημαϊκούς ε, κλπ για συζητήσεις που διεξάγονται πάνω στο θέμα αυτό. Τώρα άκουσα για το κέρα της Αφρικής, είναι μια περιοχή την οποία παρακολουθώ εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα και θα πρέπει να υπάρχει κάποιο ειδικό απεσταλμένο προκειμένου να βοηθήσει στην καταπολέμηση τη πειρατεία κλπ. Αλλά η ομάδα μου είναι αντίθετη με το να αποστέλλονται κάποιοι ειδικοί απεσταλμένοι σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα. Ευχαριστώ. Κύριε Τάνοκ, ζήτησε να παρέμβει και η κυρία Μπράντενερ. Έχετε το λόγο. Εγώ έχω μια σύντομη πρακτική ερώτηση. Δεν μου έχει, μου έχει ακόμα απαντήσει κανείς, αλλά για την αμοιβή του διπλού, του διπλού τι θα κάνουν, θα λάβουν το ένα από τα δύο. Αυτό είναι ίσως μια ερώτηση που μάλλον ο κύριος Παπόφσκι θα πρέπει να απαντήσει και όχι ο κύριος Άντεμπάρα. Απαντήστε εσείς στον Τάνοκο, στο εν μεταξύ ο κύριος Παπόφσκι να σκεφτεί την απάντηση. Στον Τάνοκ να απαντήσετε. Ναι. Τα επιχειρήματα υπέρ των περιφερειακών ευρωπαϊκών απεσταλμένων είναι περισσότερα από ότι υπέρ των ε, πεσταλμένων αναχώρα. Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Αν δούμε την Βοσνία Ζεγοβίνη, το Κοσφοπέδιο που αναφέρθηκαν, η πρόθεση είναι αυτή, αλλά η κατάσταση επιτόπου δεν βοηθά ώστε να υπάρχει ε, κάποιος ε, ειδικός απεσταλμένος ο οποίος να είναι πρώτα ο αρχηγός της αποστολής εκεί. Ε, θα πρέπει αυτή η μετάβαση να γίνει και φαντάζομαι ότι ε, οι προτάσεις της είπα της εκπροσώπου ε, για την σταδιακή, το σταδιακό phase out ε, αφορούσε τέτοιου είδους εντολές. Ε, όμως περιλαμβάνονταν και δύο περιφερειακές εντολές ε, που δεν, ε, όπου δεν έστεκαν τα ίδια επιχειρήματα. Όταν ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας μπορεί να καλύψει τη σύγκρουση θα πρέπει αυτό να το αναλάβει. Και το λέω αυτό με προσοχή διότι υπάρχουν χώρες όπου ο ειδικό απεσταλμένος αναχώρα έχει πλήρη, πλήρη απασχόληση το να, να λάβει ένας επικεφαλής αντιπροσωπείας και αυτό, σε ορισμένε χώρε λοιπόν, ίσω να είναι περιβολικά πολύ όγκο δουλειά. Αλλά βέβαια και η Λέδη Άστον έχει δύο δουλειέ να κάνει και τι κάνει. Δεν είναι το κεντρικό επιχείρημα. Πρέπει προσεκτικά να γίνει η μετάβαση. Σα ευχαριστώ. Δόκτωρα Άδεπερ, ο δόκτωρ Ποπόφσκι απαντήσει ίσως το ερώτημα ποιος πληρώνει και πόσα. Να σας δώσω την καλύτερη δυνατή εκτίμηση, αλλά, γιατί δεν είμαι αρμόδιος για το θέμα. Πόσο γνωρίζω, αυτοί που είναι επικεφαλής των ευρωπαϊκών αντιπροσωπιών που έχουν και αναλάβει τώρα να είναι ειδικοί επεσταλμένοι πληρώνονται ω επικεφαλής των αντιπροσωπιών. Μπορώ να το ελέγξω γιατί δεν είμαι πολύ τα σίγουρο. Έχουμε και άλλου. Στη Βοσνία, για παράδειγμα, ειδικού επεσταλμένους, όπου το διπλό έργο είναι διαφορετικής φάσης ε, φύση, συγγνώμη, γιατί έχουν και διεθνή λειτουργία, όπως ε, το, ε, έχουν αναλάβει το γραφείο του υπό εκπροσώπου και γι' αυτό και παίρνουν και έναν μισθό του ΙΕ. Θα το ελέγξω ξανά στη διοίκηση και θα επανέλθω. Θα δώσω την απάντηση στην κυρία Κοιτάξτε, εγώ ρώτησα αυτή την ερώτηση γιατί πολλοί δημοσιογράφοι ασχολούνται με το θέμα. Bene, lo facciamo per iscritto. <laughs> Ωραία, λοιπόν, γραπτό θα σα απαντήσουμε. Ωραία, λοιπόν, να κλείσουμε τη συζήτηση εδώ. Ευχαριστώ όλου όσου παρενέβησαν, του συναδέλφου. Το θέμα είναι ενδιαφέρον, χρήσιμο που το συζητήσαμε. Έχουμε αρμοδιότητα διαβούλευση και όχι συναπόφαση ε, εδώ, αλλά... Καλό είναι να γνωρίζουμε τι συμβαίνει και να δώσουμε και τις δικές μας προτάσεις εκτός από τα σχόλια που ακούσαμε. Μέχρι τις 11 και 4 το διακόπτουμε τώρα, οπότε θα γίνει η ανταλλαγή απόψεων με τον David O'Sullivan και τον πρέσβη Χίσοφ σχετικά με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τη Νέα Συμφωνία ΕΕ Ρωσίας.

Please, colleague, sit down. The... Our... Καθίστε, συνάδελφοι, παρακαλώ. Ο καλεσμένος μας είναι εντός αιθούσης και έχουμε πολύ φορτωμένη μερίσια διάταξη. Και έχουμε ήδη αργήσει πέντε λεπτά. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων ε, σχετικά με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τη Νέα Συμφωνία Ένωσης Ρωσίας. Γνωρίζετε ότι το φθινόπωρο του 2010 έγιναν δύο γύροι διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία. Και είναι λοιπόν σκόπε με μια ανταλλαγή απόψεων για να ενημερωθούμε ως Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων όπως προβλέπετε και από την πολιτική συμφωνία ανάμεσα στον είπατε εκπρόσωπο και την εφαρμογή του Συνθήκη τη Λισαβόνα, όπου εμπλέκει το κοινοβουλίο μα σε αυτή την υπόθεση. Δίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Ντέιβιντ Σάλεβαν που αντιπροσωπεύει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον πρέσβη Χιζόφ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω, καθώς πρόκειται για την πρώτη μου εμφάνιση ενώπιον της Επιτροπής σας υπό τη σημερινή μου ιδιότητα, τη νέα μου ιδιότητα, να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Γνωρίζετε την μεγάλη ε, δέσμευση της ΥΠΑ της εκπροσώπου να έχει στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Και Είτε πρόκειται για διοικητικά και οικονομικά ζητήματα, είτε πρόκειται για θέματα πολιτικής φύσης, όπως σήμερα το πρωί. Είμαι στη διάθεση της Επιτροπής σας για οποιασδήποτε πληροφορίες και διευκρινήσεις χρειάζεστε. Και προσβλέπω στην καλή συνεργασία με την Επιτροπή σας, όπως ε, είχα εξάλλου και με την Επιτροπή ΙΝΤΑ, όταν ήμουν υπεύθυνο για το εμπόριο, στην προηγούμενη μου ζωή ε, στην προηγούμενη μου ιδιότητα. Και τελευταία φορά που εγώ και ο πρέσβης συναντηθήκαμε ήταν ε, στην ε, τέλος των διαπραγματεύσεων στις οποίες συμπροέδρευα ε, τότε μαζί του ως υπεύθυνο της Ρέλεξ. Ένα λεπτό μετά από τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου άλλαξα ιδιότητα και τώρα είμαι πρόσωπος της υπηρεσία Εξωτερικές δράσεις. Θα ήθελα να σα ενημερώσω και εξάλλου και ο πρέσβη θα σας πει ποιες είναι οι δικέ του προεπτικοί για αυτές τις διαπραγματεύσει. και πρόκειται για δυόμιση έτη διαπραγματεύσεων πολύ σημαντικών και για μια πολύ σημαντική συμφωνία. Όπω ξέρετε ξεκίνησαν όλα αυτά το 2008, έχουμε δύο δεκαγύρου διαπραγματεύσεων όπω θα θυμάστε και θα έλεγα ότι υπάρχουν καλά νέα και λιγότερο καλά νέα. Τα καλά νέα ότι έχει γίνει πρόοδος, πολύ πρόοδος και σε αυτά θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω πως τα λιγότερο καλά νέα είναι ότι ίσως να μην μπορέσαμε να προχωρήσουμε τόσο και τόσο γρήγορα στον τομέα των εμπορίων και των επενδύσεων όσο θα θέλαμε. Και θα θέλαμε ο τομέα αυτός να προλάβει και τις υπόλοιπες διαπραγματεύσεις, τους υπόλοιπους τομείς, ώστε να μπορέσουμε να, φτάσουμε, να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις. Όπως γνωρίζετε, στόχος μας είναι καταρχήν θέλουμε να έχουμε ισχυρή και φιλόδοξη και καθολική εταιρική σχέση και συμφωνία συν Plus που θα δώσει μεγαλύτερη αξία στην ισχύουσα συμφωνία, περισσότερα να πετύχουμε δηλαδή και όχι λιγότερα με βάση την PCA και τους κοινού χώρους και εργαζόμαστε για την ενημέρωση και τη συμπλήρωση της ισχύουσα, των ισχυουσών ε, υποχρεώσεων σύμφωνα με την ε, Συμφωνία εταιρική ε, Σχέσης. Ένα θέμα το οποίο γνωρίζω καλά από τις προηγούμενες μου είναι αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι μια νέα συμφωνία χωρίς ε, ουσιαστικό θεμελιώδες εμπόριο και, συναλλαγό, και συναλλαγές συμπεριλαμβανομένου σε τις ενέργειες δεν θα ήταν ε, υποδεκτή επιλογή για μας και είμαι ευχαριστημένη για, ευχαριστημένος για τον πρόοδο που έχει σημειώσει η Ρώσα για την προσχώρηση στον ΠΟΕ ε, και ελπίζω πως έτσι θα προχωρήσει και στις πολυμερείς συζητήσεις η κατάσταση σύντομα. Βέβαια παραμένει ένα ανοιχτό θέμα, δηλαδή οι συγκεκριμένες επιπτώσεις της δημιουργίας της Τελωνιακής Ένωσης για τις διμερείς μας εμπορικές σχέσεις αλλά υποστηρίζουμε την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλα τα μέρη ώστε αυτό να επιτευχθεί όσο γίνεται πιο σύντομα. Έπειτα κάτι ακόμα το οποίο υποθέτουμε βεβαίω είναι ότι η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών θα αποτελέσουν ε, βασικό στοιχείο αυτή τη συμφωνία. Ένα στοιχείο το οποίο η παραβίαση θα αποτελούσε βάση για μονομερή αναστολή τη συμφωνία. Αν ε, συνέβαινε κάτι τέτοιο για μα, τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στην καρδιά των σχέσεών μα και, και πρέπει αναλόγω να αντιμετωπίζονται και στη νέα συμφωνία. Και είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι στην ισχύουσα συμφωνία ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και της ε, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 και δεν πρόκειται να χαμηλώσουν οι προδιαγραφές ε, ως προς αυτό στη νέα συμφωνία. Δεν θέλω να καταναλώσω χρόνο. Είμαι λεπτομέρειες αλλά να σας αναφέρω κάπως τι διαπραγματεύσεις που γίνονται σε τέσσερις ομάδες εργασίας. Πολιτικός διάλογος για την εξωτερική ασφάλεια. Δεύτερον, ελευθερία, δικαιοσύνη και ασφάλεια. Τέταρτον, οικονομικά θέματα. Και τέταρτον, έρευνα, παιδεία και πολιτισμός. Να σας δώσω μια γεύση για το τι συμβαίνει σε αυτές τις ομάδες. Όταν συνεδριάσαμε το Δεκέμβριο, ο πρέσβης και εγώ μπορέσαμε να σημειώσουμε πρόοδο στο τομέα του πολιτικού διαλόγου της εξωτερικής ασφάλειας και της ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η σύνταξη του κειμένου για τον πολιτικό διάλογο και την εξωτερική ασφάλεια έχει προχωρήσει. Τα θέματα για τα μικρά όπλα ε, και για την πολιτική προστασία έχουν προσωρινά ολοκληρωθούν, ε, ολοκληρωθεί και κοντεύουμε να ολοκληρώσουμε και τις διαπραγματεύσεις για τα ε, όπλα μαζικής καταστροφής. Χρειάζεται όμως κάποιο ξεκαθάρισμα. Υπάρχουν περισσότερες δυσκολίες για τις βασικές αρχές συνεργασίας στον τομέα αυτό. Θα θέλαμε να υπάρξει μια παραπομπή στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ των βασικών αρχών μαζί με τον ε, σεβασμό για το κράτος δικαιού. πρέπει να σα εξηγήσει φυσικά τη θέση του, αλλά θα έλεγα ότι η Ρωσία έχει επιφυλάξει σε σχέση με το αν η δημοκρατία είναι μια αρχή και, και θεωρεί ότι η αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι υπερβολικά πολυάριθμη μέσα στο κείμενο. Τελικά, ίσως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για περιοχές ε, που είναι κοντινές, στη, ε, κοντινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ρωσική ε, Ομοσπονδία. Η Ρωσία θέλει να συνοδευτεί η λέξη ασφάλεια από τις λέξεις ισότιμη και, μη, και, και διαφυσβήτητη ασφάλεια ε, είναι λέξεις στις οποίες μπορούν να συνοδεύουν ένα, τη λέξη ασφάλεια σε ένα νομικό κείμενο. Σχετική πρόοδος έχει συμβιωθεί στο ομάδα εργασίας ελευθερία, ε, δικαιοσύνη ε, και ασφάλεια έχουν ολοκληρωθεί οι διατάξεις ε, για το οργανωμένο έγκλημα καθώς και τη διαχείριση των συνόρων αλλά παραμένουν διαφορές ε, όσον αφορά το άσυλο, τη μετακίνηση ανθρώπων και τη δικαστική συνεργασία καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα αναφερθούμε στις γενικές αρχές του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ήδη σας ανέφερα. Υπάρχει επίσης το θέμα της σύνδεσης ανάμεσα σε, μια, σε αυτή τη συμφωνία και την πρόοδο για το θέμα των θεωρήσεων που θεωρούμε πως είναι κάπως διαφορετικό γιατί υπάρχει διαφορετική οδός που έχει συμφωνηθεί εδώ. Πάντως είναι σαφές ότι όποια πρόοδο και αν σημειωθεί εκεί θα αντικατοπτριστεί και στην συμφωνία όταν αυτή ολοκληρωθεί. Για το θέμα της οικονομικής συνεργασίας έχουμε και εκεί σημειώσει πρόοδο Έχουμε κλείσει περίπου 11 κεφάλαια, δεν θα σας τα παριθμίσω, αλλά καλύπτουν τη στατιστική, το διάστημα, τον τουρισμό, την ανάπτυξη της υπαίθρου και ούτω καθεξής. Και συνεχίζεται η σύνταξη για τέσσερα ακόμα ε, κεφάλαια, καθώς και για περισσότερα και άρθρα συνεργασίας που θα τεθούν επιτάπητος από τη στιγμή που θα έχουμε μια σαφή εικόνα για τις οριζόντιες διατάξεις για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Και εδώ έρχομαι στον τομέα που μας ε, δημιουργεί τις περισσότερες δυσκολίες για την ώρα. Όταν δηλαδή πέρσι ο κύριος Μιγκαρέλ ήταν εδώ εξ ονομά της Επιτροπής τότε. Τον Ιούνιο σας ενημερώσαμε ότι θα καταθέταμε το πρώτο κομμάτι των διατάξεων περί εμπορίου και επενδύσεων αφορούσε τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο, δικαιώματα πνευματικά, εμπόριο αγαθών, θέματα διαφάνειας κτλ. Τώρα έχουν όντω στεθεί στην ε, Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων από τον Ιούλιο του 2010. Δεν έχουμε ακόμα λάβει το είδο τη ε, ουσιαστική ε, αντίδραση που ελπίζαμε από του Ρώσου εταίρου μα, αλλά στην ουσία έχουμε κάνει μόνο μια αρχική ανταλλαγή απόψεων. Συμφωνήσαμε για τον 11ο γύρο διαπραγματεύσεων να δημιουργήσουμε μια ομάδα συντακτική που θα αποτελείται από εμπειρογνώμονε στα θέματα αυτά, ώστε να προχωρήσουν λεπτομέρειε. Η συντακτική ομάδα έχει συναντηθεί δύο φορέ πριν από τον 11ο γύρο, αλλά ειλικρινά δεν έχει σημειωθεί πολύ μεγάλη πρόοδο και φοβούμε ότι θα πρέπει να πω το ίδιο και για την τελευταία συνεδρίαση τη ομάδα εργασία για τα οικονομικά ζητήματα που έγινε στι Δεκεμβρίου. Είναι μια, ένας τομέας που δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά στις Ε, πιστεύω ότι ο πρέσβης και εγώ συμφωνήσαμε να εντείνουμε τις προσπαθίες μας στον τομέα αυτό. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσουμε πόρους και ενέργεια για τις διαπραγματεύσεις ε, των διατάξεων για το εμπόριο και τις επενδύσεις και θα επανέλθουμε στις πιο ε, προηγμένες ομάδες μετά. Έχουμε προγραμματίσει συνεδρίαση της ομάδας αυτής της συντακτικής στις 4 Φεβρουαρίου. Ε, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Δύο τελευταίες παρατηρήσεις. Έχει υπάρξει πρόοδος για την παιδεία και τον πολιτισμό. Το κεφάλαιο για την παιδεία, την κατάρτιση, τον αθλητισμό και την νεότητα έχει προσωρινώς κλείσει. Για την πολιτισμό έχουμε κάποια διαφορά απόψεων για το πώς θα μιλήσουμε για τα θέματα για την πολιτιστική διαφορά και για το θέμα των πολιτιστικών αγαθών έπειτα και θα συνεχίσουμε να διερευνούμε λύσεις εδώ. Τέλος, δύο λόγια για το θέμα της έρευνας. Έχουμε στείλει επισήμω πρόσκληση στη ρωσική πλευρά για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει για τη σύνδεση τη Ρωσία με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Έρευνα, ε, πρόγραμμα πλαίσιο μάλλον, ε, που έχει ζητήσει από το 2008. Το έχουμε αυτό βάλει στο πλαίσιο τη Νέα Συμφωνία. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε επίσημη απάντηση στην επίσημη μα πρόσκληση, αλλά υπήρξε επιστολή από τον ε, Υπουργό Φωσέγκο που υποδεικνύει ότι η ρωσική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να δεχτεί την πρόσκληση για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για τη Νέα Συμφωνία όσο γίνεται πιο σύντομα. Οπότε, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, νομίζω πως... Ε, πολλά θετικά στοιχεία υπάρχουν στα όσα σας ανέφερα, έχει γίνει πρόοδος, αλλά είναι λίγο άνηση. Και πιστεύω ότι θα πρέπει τώρα να βάλουμε λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια στον τομέα των εμπορίων και των επενδύσεων, ώστε να είναι ισορροπημένες οι διαπραγματεύσει που θα προχωρούν σε όλα τα μέτωπα που είναι σημαντικά για μας ταυτόχρονα. Φυσικά είμαστε προσιλωμένοι στην, στην αίσια έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων όπως και ο πρέσβης ε, και πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε τώρα μια επιπλέον προσπάθεια στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, δόκτωρα ο Σάλιμπαν, και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον ε, ε, πρέσβη Χίσοφ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής ε, της Ρωσικής ε, Αντιπροσωπείας ε, για τη Συμφωνία. Χθες ε, τηρήσαμε ενό λεπτού στη γη για τα θύματα του Ρωσικού αεροδρομίου. Ε, σας εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας, ε, τη συμπαράστασή μας προς το ρωσικό λαό για το πένθος σας αυτή η βάρβαρη πράξη μας οδηγεί νομίζω στο να νιώθουμε ακόμα πιο δυνατοί ώστε να συμβάλλουμε και εμείς στην αναζήτηση μιας πολιτικής λύσης για να αντιμετωπιστούν οι σειράξεις που πλήττουν τον Κάφκασο. Βεβαίως καταδικάζουμε αυτές τις φρικόδεις και βίες πράξεις. Ε, κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συλληπιτήριά σας και για την συμπόνια που επιδείξατε σε αυτή την ε, βάρβαρη επίθεση που δέχτηκε το αεροδρόμιο της ε, Μόσχας εχθές ή προχθές. Ευχαριστώ επίσης και για την ευκαιρία που μου δίνετε να συναντηθώ με τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω το δικό μας το όραμα για τη νέα συμφωνία που πρόκειται να συναυτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω τον κύριο Σάλεβαν, τον συνδιαπραγματευτή μου, αν μου επιτρέπετε να τον χαρακτηρίσω έτσι, για ε, την επιτυχία και για τα δύο, και για την επιτυχία και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Κανείς δεν περίμενε ότι θα πρόκειται για μια εύκολη διαδικασία. Με λίγα λόγια θα μου επιτρέψετε να σας ε, σκιαγραφίσω το ιστορικό όλων αυτών των διαπραγματεύσεων. Η ιδέα που υπάρχει για τη νέα συμφωνία, νέα συμφωνία είναι βέβαια προσωρινός ο τίτλος. Θα επανέλθουμε ε, στον τίτλο της ε, συμφωνίας από τη στιγμή που θα λάβει τελική μορφή το κείμενο. Η ιδέα λοιπόν που διατρέχει όλο αυτό το σκεπτικό είναι ότι η νέα συμφωνία θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα συμφωνία ε, συνεργασίας ε, και εταιρική σχέσης ε, που ολοκληρώθηκε το 1997 και εξακολουθεί βέβαια να ισχύει ανανεούμενη αυτόματα σε αιτήσια βάση. Μέχρι βέβαια μία από τις δύο πλευρές εκφράσει την επιθυμία της να πάυσει να ισχύει η συμφωνία αυτή. Πριν λοιπόν αποφασίσουμε, πριν οι ηγέτες μας αποφασίσουν να ε, ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, εμείς μελετήσαμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις που είχαμε, όπως επίσης και την εμπειρία που έχει αποκομίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλους τρίτους εταίρους, Ηνωμένε Πολιτείε, Ιαπωνία, Κίνα, Νορβηγία, Ελβετία. Καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η καλύτερη λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία είναι να υπάρξει μια νέα περιεκτική ευρεία συμφωνία. Και αυτό αποφασίστηκε το 2005 σε μια συνάντηση κορφή στο Λονδίνο. Η ρωσική κυβέρνηση αποφάσισε να είμαι εγώ ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων. Αυτό αποφασίστηκε τον Νοέμβριο του 2005. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάστηκε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να πράξει και εκείνη το ίδιο. Κατόπιν τούτου το μόνο που κατορθώσαμε ήταν να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις τον Ιούλιο του 2008. Η όλη ιδέα πίσω από αυτή τη νέα ευρεία συμφωνία είναι νομίζω κατανοητή. Αν πάμε πίσω στο 94 θα καταλάβετε πολύ εύκολα πόσο άλλαξε έκτοτε η Ρωσία αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τομείς ε, συνεργασίας που δεν καλύπτονται από αυτή τη συμφωνία. Παραδείγματος χάρη συνεργασία ε, στον τομέα της ΚΕΠΑ δεν υπήρχε ΚΕΠΑ ε, το 1994 και σε πολλούς άλλους τομείς υπήρξαν αλλαγές. Ας πούμε, αυξάνει όλο και περισσότερο το εύρος της ε, συνεργασίας. Πώς θα, ποιος θα πίστευε ποτέ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία από κοινού θα ε, προσπάθουν να καταπολεμήσουν την δεκαετία του 90 την πειρατεία έξω από τις ακτές της Σομαλίας. Ο στόχος της νέας συμφωνίας είναι να γίνει ένα ποιοτικό βήμα προς τα εμπρός, μια ενισχυμένη νομική βάση ε, που θα δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες σε αυτή τη συμφωνία. Η συμφωνία θα πρέπει να είναι ρηξικέλευτη, ε, διορατική, ε, να αναθεωρεί τις στρατηγικές μας σχέσεις. Βεβαίως θα πρέπει να είναι ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο και υπάρχει για μας κι άλλος ένας λόγος γιατί εμφανιζόμαστε σε αυτή την Επιτροπή. Διότι εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού με το ε, Ρωσικό Κοινοβούλιο να επικυρώσουν το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας. Πριν λοιπόν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις τον Ιούνιο του 2008 οι επικεφαλής της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη αυτών των διαπραγματεύσεων και ανέφεραν ότι η νέα συμφωνία θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τομείς των σχέσεων ε, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικούς ε, χάρτες πορείας και παράλληλα έδωσαν και τη δυνατότητα να αναπτυχθούν περαιτέρω τομεακές συμφωνίες που καλύπτουν διάφορους τομείς της ε, συνεργασίας. Μιλάμε λοιπόν για μια συμφωνία που θα είναι ευρεία, αλλά όσο ευρεία και αν είναι, οι δύο πλευρές δεν έχουν ως στόχο να καταλήξουν σε ένα κείμενο που θα καλύπτει τα πάντα. Εγώ θεωρώ περισσότερο ότι είναι ένα έγγραφο σκελετός ε, στο οποίο θα προστίθενται και άλλες τομεακές συμφωνίες. Και θα υπάρχει βέβαια και ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που ακόμα δεν έχουμε αρχίσει να το συζητάμε ε, σχετικά με τις ε, κατάλληλες ε, θεσμικές πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν για να λειτουργεί εύρυθμα αυτή η συμφωνία. Το αποτέλεσμα λοιπόν των 12 γύρων διαπραγματεύσεων, κατά τη γνώμη μου, είναι θετικό. Κανείς δεν περίμενε όπως σας είπα ότι θα ήταν μια εύκολη διαδικασία, αλλά και κανείς δεν περίμενε ότι ε, η διαδικασία θα προχωρήσει με ταχύ ρυθμό. Είναι λοιπόν μια διαδικασία η οποία επηρεάζεται ε, δυστυχώς και από μια τεχνητή ημερομηνία καταληκτική. Και μας ενδιαφέρει περισσότερο η ποιότητα και όχι τόσο το χρονοδιάγραμμα από ό,τι φαίνεται. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ήδη ανέφερε ο Ντέιβιτ σχετικά με τα αποτελέσματα των τεσσάρων ομάδων εργασίας. Πράγματι, τα θέματα του εμπορίου αποδείχτηκε ότι ήταν ένας από τους δυσκολότερους τομείς. Επίσης, όσον αφορά στον ορισμό των ορίων ανάμεσα στη βασική συμφωνία και την προτιμησιακή δεύτερη συμφωνία ε, αυτά τα όρια θα ακολουθήσουν, η χάραξη των ορίων. Επίσης, ε, εμείς ξεκινήσαμε από την παραδοχή ότι αυτή η νέα βασική συμφωνία θα συναυτεί ανάμεσα σε μέλη του ΠΟΕ. Η διαδικασία ένταξης των ΠΟΕ είναι βέβαια μια ξεχωριστή διαπραγμάτευση και αυτή μπορεί να κλείσει μετά από 17 χρόνια. Έχει ήδη κλείσει 17. Αυτό είναι ρεκόρ Guinness. Η δική μας η διαδικασία είναι ακόμα πιο χρονοβόρα από αυτή των Κινέζων. Αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύουμε ότι τώρα πια μήνες μόνο λείπουν και όχι χρόνια μέχρι να ε, ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής μας στον ΠΟΕ και έχω τη χαρά να σας ανακοινώσω ότι το μνημόνιο κατανόησης το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 7 Δεκεμβρίου του 2010 και επικυρώθηκε ε, την ίδια μέρα στη συνάντηση κορυφής αυτό περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία των ε, διμερών διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας για την ένταξη στον ΠΟΕ. Το κακό είναι ότι ο ΠΟΕ δεν περιλαμβάνει μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ρωσία, έχει και πολλά άλλα μέλη. πάση περιπτώσει, εμείς ε, προτιθέμεθα ε, να δώσουμε μια τελική μορφή σε αυτή τη συμφωνία και στη διαδικασία μάλλον το συντομότερο δυνατόν. Κατά την άποψή μας, εκείνο που είναι απαραίτητο για να υπάρχει σταθερή πρόοδος είναι ίσως όχι η επιτάχυνση αλλά περισσότερο ε, σταθερή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και τα δύο μέρη είναι έτοιμα και έχουν και την απαραίτητη πολιτική βούληση για σύναψη συμβιβασμών. Ε, κατά την άποψή μου, στο εγγύς μέλλον, η διαπραγματευτική εντολή από την, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, μετατεθεί από την Επιτροπή προς την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και αν κάνω λάθος, παρακαλώ, διορθώστε με. Ελπίζω ότι η διαπραγματική, διαπραγματευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει το απαραίτητο περιθώριο ελιγμών για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. Μάλιστα, ένα από τα στοιχεία που παρακόλλησαν μέχρι τώρα την διαπραγματευτική διαδικασία ήταν το γεγονός ότι από τότε που ξεκινήσαμε, ο Ντέιβιτ είναι ο τέταρτος συνομιλητής μου στις διαπραγματεύσεις. Έναν ένα τους χάνω. Ελπίζω αυτός τουλάχιστον να μου μείνει. Δεύτερον, νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε βήματα που θα οδηγούσαν ενδεχομένως στο ε, να σπάσει η συμφωνία. Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουμε στο όραμα της νέας συμφωνίας που όπως σας είπα ε, θα είναι ευρεία. Δεν πρέπει λοιπόν να δημιουργούμε προβλήματα ούτε στη μία πλευρά ούτε στην άλλη. Να μην δημιουργούμε προσκόμματα στις διαπραγματεύσεις. Γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό είναι αλυσίδα, θα προκύψουν και άλλες δυσκολίες. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή τη φιλόδοξη συμφωνία η οποία όπως σας είπα ε, θα είναι στο σωστό επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία κάτω από μέσο μακροπρόθεσμη προοπτική. Σας ευχαριστώ. Και εμείς, κύριε Πρέσβη, ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση με την πρώτη παρέμβαση που είναι ο συγητής μας για τη ε, συμφωνία αυτή. Ο κύριος Σεβερίν, παρακαλώ τρία λεπτά. Μόνο ότι έχω λίγο χρόνο στη διάθεσή μου, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και την θλίψη μου στον ρωσικό λαό που έζησε αυτή την βαρβαρότητα της τρομοκρατίας και ο κύριος πρέσβης αναφίβολα θα διαβιβάσει τα συλληπιτήριά μας στους συμπολίτε του. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω και του δύο συνομιλητέ για τη δουλειά που έχουν ήδη κάνει αλλά και για τι προφορίε που μα δίνουν. Σίγουρα ήταν πολλέ οι προφορίε που ακούσαμε και το θεωρώ ως ε, μια διάφανη, διάφανη προφόρηση, για τις διάφανες ε, διαπραγματεύσεις, ε, κάτι το οποίο μας επιτρέψει να αντιδράσουμε αποτελεσματικά. Επίσης ε, θα ήθελα να πω ότι τίποτα σε αυτή τη συμφωνία, τίποτα σε αυτή τις διαπραγματεύσεις δεν είναι καθαρά τεχνικό, όλα τα ζητήματα είναι πολιτικής φύσης και τίποτα δεν είναι μια απλή διαδικασία σε σχέση με τις ε, σχέσεις που έχουμε με τη Σοβιετική Ένωση, αλλά είναι, καταβάλλονται επειδή τις προσπάθειες ώστε να προετοιμάσουμε ένα στρατηγικό πλαίσιο και τις κατάλληλες νομικές βάσεις για μια μακροχρόνια ε, σχέση σε εμπορικό και πολιτικό επίπεδο με τη Ρωσία. Να πω επίσης πως η νέα συμφωνία θα περιέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο και θα συμπεριλαμβάνει επίσης τις νομικά δεσμευτικές δεσμεύσεις της, των δύο μερών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία κλπ, εξωτερική πολιτική, διάλογο, καταπολέμηση τρομοκρατία, ε, Αφγανιστάν, Ιράν, σταθερότητα στην Κεντρική Ασία, την επίλυση ε, σειράξεων, ε, θέματα ελευθερίας, δικαιοσύνης, διευκολύνσεις θεωρήσεων, διακίνηση προσώπων, οικονομική συνεργασία και την συμμετοχή της ε, Ρωσίας στον ΠΟΕ, θέματα ενέργειας κλπ. Προκειμένου να πετύχουμε σε όλα αυτά, θεωρώ ότι πρέπει να ε, επικρατεί το κλίμα εμπιστοσύνη ε, κάποιες αδυναμίες θα καταστήσουν τα πράγματα πιο περίπλοκα και δύσκολα και ναι, πω τον κύριο Σάλβαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει σαφείς εγγύησεις προς τη Ρωσία και να την πείσει ότι είναι καλύτερο να έχει στενές και ισχυρές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση μελώντης και όχι με τα επιμέρους κράτη της ε, και θα πρέπει να βλέπουμε τη Ρωσία ως έναν αξιόπιστο εταίρο. Τώρα, μερικές πολύ σύντομε ερωτήσει για την ε, ένταξη στον ΠΟΕ. Φυσικά τα διμερεί θέματα μπορεί να έχουν επιληθεί, αλλά υπάρχει κίνδυνος ε, κάποια άλλα κράτη-μέλη να παρεύουν ε, με τρόπο λιγότερο θετικό στην διαδικασία. Η προσχώρηση της Ρωσίας δεν είναι μόνο προς όφελος της Ρωσίας, αλλά και προς όφελος της Ευρώπης. Ίσως κύριε Πρέσβη θα μπορούσατε να μας πείτε πώς είναι δυνατόν να βοηθήσουμε την όλη διαδικασία χρησιμοποιώντα τι δικέ μα ε, σχέσει και επαφέ με τρίτε χώρε. Θα ε, φτάσω τώρα στο ζήτημα των θεωρήσεων. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα και ίσω ο κύριο Πρέβη θα μπορούσε να μα δώσει περισσότερε λεπτομέρειε για πράγματα τα οποία δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, διότι φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλε καθυστερήσει. Και τέλο, δεν μιλήσατε πολύ για τον εξυγχρονισμό τι η Ρωσία προσβλέπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα εξεχρονισμού. Νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία και για τη Ρωσία αλλά και για μας. Και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τον, τον εξυγχρονισμό που είναι μια έννοια πολύπλευρη και πολυμερής. Ευχαριστώ. Κύριε Σεβερίν, το λόγο έχει ο κύριος Σάλα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Σάλιβαν για την ε, παρουσία του και να τον συγχαρώ επί τη αναλήψη των νέων καθηκόντων ε, στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Νομίζω ότι η μέχρι τούδε θητεία του και η θέσεις που κάλυψε μέχρι τώρα μας ε, κάνουν να πιστεύουμε ότι θα βάλει τάξη πράγματα. Ευχαριστώ επίσης τον Ρώσο Πρέσβη εξ ονόματος του ΕΛΚ να του εκφράσω την ελεγγύη μου όπως είπε και ο Πρόεδρος που εξάλλου μας ζήτησε να κάνουμε, τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Συμφωνώ με την εισαγωγή του Ρώσου Πρέσβη ότι δηλαδή αυτή η συμφωνία θα πρέπει να αποτελέσει μια, ένα ποιοτικό άλμα στη σχέση μας. Θεωρώ ότι ως σημαντική εταίρη αυτός αυτή η συμφωνία πρέπει να στηρίζεται σε αρχές και άξιες. Νομίζω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να είναι ε, μια ρήτρα βασική στην όλη συμφωνία. Θα πρέπει να είναι αμοιβαία αυτή η απέτηση και γι' αυτό με ιδιαίτερη ικανοποίηση άκουσα τις δηλώσεις του κ. Σάλιβαν και εντάχει δύο ερωτήσεις. Το ζήτημα της, ε, των επενδύσεων και του εμπορίου, το συγκεκριμένο και καθυστέρησή του. Το... Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω κάποιες ε, εξηγήσεις γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Ο κύριος Σεβερίνος, συγητή, ε, μα είπε ότι σε αυτή τη συμφωνία όλα έχουν πολιτική, είναι πολιτικής φύσης. Αλλά να αναρωτιέμαι πώς το πλαίσιο τη νέα στρατηγική ε, για τον σύμφωνο για το Ατλαντικό Σύμφωνο θα μπορούσε να επηρεάσει λοιπόν τα διάφορα κεφάλαια τα οποία αφορούν στο το κομμάτι της ασφάλειας. Κύριε Σάλιβαν, μιλήσατε για γειτονικέ περιοχές και όχι για γείτονες. Εμείς έχουμε μια πολιτική γειτονία που έχει ε, μια συγκεκριμένη ορολογία. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε κάτι σχετικά με την εμπειρία αναφέρθηκε σε αυτό ο κύριος Σιγητής, ε, δια της ε, προξενικές θεωρήσεις. Λοιπόν, ποια είναι η εμπειρία λοιπόν, που έχουμε αποκτήσει, ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, αυτά μας λένε ότι οι Ρώσοι πολίτες έχουν στήσει το δι, δι, θεωρήσεις από ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Υπάρχουν και άλλες πτυχές κύριε Πρόεδρε, δεν έχω χρόνο στην διάθεσή μου. Η κρίση στην Γεωργία και το πώς έχουν διαπραγματεύσεις ε, πάνω στο θέμα αυτό. Ελπίζουμε ότι το έμπειρο χέρι του κυρίου Σάλιβαν θα μπορέσει να καθοδηγήσει τις διαπραγματεύσεις αυτές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο Μανδρόη, ε, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου σε μια πρώτη φάση να πω πως συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπατε εσείς Πρόεδρε αλλά και ο συνάδελφος μου Σάλα Φράγκα προκειμένου για την ε, Συμφωνία τελικής Σχέσης ε, θεωρώ ότι σε μια πρώτη φάση έχουμε έναν κοινό χώρο, μετά ε, δημιουργήσαμε την εταιρική σχέση για τον εξυγχρονισμό και τώρα μας, ε, συνεχίζει να μας απασχολεί αυτό το ζήτημα της Συμφωνίας Συντηρικής Σχέσης. Νομίζω λοιπόν ότι τόσο αυτό το ζήτημα όσο και η ατζέντα για τον εξυγχρονισμό μας παρεμπόδιζαν στο να προχωρήσουμε περαιτέρω στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Είναι αυτό, είναι κάτι το οποίο πράγματι με λυπεί, διότι αυτή η συμφωνία εσωτερική σχέση και συνεργασία είναι σημαντική όχι μόνο για μας αλλά και για τη Ρωσία. Να προσθέσω επίση και κάτι ακόμα. Θεωρώ πως ε, οι απόψεις μας ε, μπορεί να διαφέρουν σε κάποια θέματα. Η Ρωσία λέει πρέπει να βιαστούμε, να προχωρήσουμε γρήγορα, αλλά εμείς ζητάμε ότι χρειάζεται να συμπεριληφθούν και κάποια άλλα στοιχεία και δι' τα εμπορικά. Έχουν την εντύπωση λοιπόν ότι απουσιάζει η αμοιβαιότητα. Άλλη μια παρατήρηση, Πρόεδρε. Τι γίνεται με τον ΠΟΕ Και κάτι ακόμα. Σε ό,τι αφορά τον ε, ναι, εξυγχρονισμό, όταν μιλάμε για εξυγχρονισμό εννοούμε και εκδημοκρατισμό. Συχνά ακούω τις επικρίσεις του Μεντβεντεύ για το κακό κλίμα που επικρατεί σε ζητήματα επενδύσεων ε, κλπ. Αλλά αν ε, βλέπουμε το τι συνέβη με τον Κοτοκόφσκι, η υπόθεση Ανίψκη, τα ζητήματα τα οποία φύγουν κάποιοι διαμαρτυρόμενοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας πείτε κάτι παραπάνω για αυτήν την ατζέντα του εξυγχρονισμού στην Ρωσία. Η ε, κυρία Γιούλαντ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα ειλικρινή συλληπιτήριά μου στην Ρωσία, στο ρωσικό λαό και την συμπαράστασή μας ε, σε όλους όσοι θρύνησαν θύματα αλλά και στο σύνολο της ε, χώρας. Έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Σάλιβαν σε σχέση με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις ε, Καλό είναι που μας είπε ότι υπάρχει πρόοδος και φυσικά η Ρωσία είναι στρατηγικός εταίρος και πρέπει να πετύχουμε αυτή την πρόοδο διότι είναι και προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ε, προείπαν και συνάδελφοι, διαπραγματεύσεις που αφορούν ε, στην εταιρική σχέση που θα στηρίζεται σε αξίες. Έχω μια ερώτηση λοιπόν που θα ήθελα να θέσω. Πώς ε, αισθάνεστε όταν διαπραγματεύεστε σε αυτό το πλαίσιο ενώ έχουμε δει πως ε, υπάρχουν διαφορετικές αξίες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό αυτών των περιπτώσεων όπως η δίκη Κοντορκόφσκι, το ζήτημα της επιρροής ε, του δικαστικού συστήματος, κάτι το οποίο έχουν καταγγείλει πολλοί διεθνείς παρατηρητές, η σύλληψη αντιφρονούντων όπως ο κ. Σεμτσόφ που δεν έκανε και τίποτα το παράνομο, δεν έδωσε λόγο προκειμένου να συλληφθεί κλπ. κλπ. Τον περασμένο μήνα στην Ολομέλεια συζητήσαμε το θέμα ενδεχόμενων κυρώσεων κατά των Ρώσων αξιωματούχων που εμπλάξαν στην υπόθεση του κυρίου Μακίνσκι και προ εβδομάδων ε, συζητήθηκε το θέμα επίσης του Κοντορκόφσκι και της δίκης του. Κύριε Σάλιβαν, λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν αλλά και οι περισσότερες εξωτερικές δράσεις μπορούν να διαπραγματεύονται μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα. Ο Ιούλαντ, ονορεύολε Σούλτς, per due minuti. will und kann mich nur den Beileidsbekundungen zu diesem schrecklichen und ε, και εγώ βεβαίως ε, θέλω να εκφράσω την αμέριστη συμπαραστασή μου ε, προς τους Ρώσους που υπέστησαν αυτές τις βίες πράξεις στο Ντομοντέντοβο, στο αεροδρόμιο της Ρωσίας. Κοιτάξτε, μας, θέλω να πω τεξί. εξής, στις διαπραγματεύσεις τσακωνόμαστε, τσακωνόμαστε πάρα πολύ και σας ερωτώ κύριε πρέσβη της Ρωσίας αυτή τη βία το κύμα βίας και την αντίδραση στη βία. Πώς θα τα αντιμετωπίσετε όταν ε, οποτεδήποτε εμφανίζεται τέτοιε πράξεις βίας, αυτομάτως το συνεπακόλουθο είναι απειλές προς τον Κάφκασο, προς χώρες του Καυκάσου. Και επίσης να πω προς τον κύριο Σάλαβαν, κοιτάξτε δεν μπορούμε και εμείς να αλλάζουμε ε, συνέχεια διαπραγματευτές, αυτό δημιουργεί ένα χάος. Από το 2009, τέλος του 2009, μιλάμε για μια συμφωνία εξυγχρονισμού με τη Ρωσία. Ε, εσείς διαπραγματεύεστε ε, παράλληλα δύο συμφωνίες που περιλαμβάνουν και μια άλλη τομεακή συμφωνία. Ε, θα συμπεριληφθούν και οι συμφωνίες ε, συνεργασίας ε, και εταιρικής σχέσης. Τι γίνεται, μήπως απλά πρόκειται για διαφορετικές επικεφαλίδες συμφωνιών. Και κάτι άλλο προς εσάς κύριε Πρέσβη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε να συσταθεί ένα φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών και να προαχθεί η συζήτηση ανάμεσα στη ΣΜΚΟ. Μάλιστα να θεσμοθετηθεί αυτός ο διάλογος. Από ρωσικής πλευράς δεν άκουσα, εσείς το στηρίζετε αυτό. Και ποιες είναι είναι οι σας ε, έτσι ώστε να συσταθεί αυτό το φόρουμ ε, κοινωνίας των πολιτών. Ευχαριστούμε τον κύριο Σούλτς, ο κύριος Τάνοκ για δύο λεπτά. Εκ μέρου ε, των Δημοκρατών Μεταρρυθμιστών σας συγχαίρω κύριε Σάλουαν και σε εσά κύριε Πρέσβη σας είπα την αμέσως συμπαράστασή μου για τα θύματα χθες στο αεροδρόμιο της Ρωσίας. Η Ρωσία είναι μια μεγάλη δύναμη και πρέπει να θεσμοθετήσει τη σχέση τη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δώσει μια συγκεκριμένη μορφή στη στρατηγική συνεργασία, να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις. Ε, η Ρωσία γνωρίζει πλέον πολύ καλύτερα τον αυξανόμενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξωτερική πολιτική. Η δική μου όμω η ομάδα εξακολουθεί να ανησυχεί όσον αφορά στο ημιαυταρχικό καθεστώς σα, όσον αφορά τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ελευθερία του τύπου, τη δικαστική εξουσία και κυρίως όσον αφορά στο να αντιμετωπιστούν, να καταδικαστούν οι ε, υπεύθυνοι για δολοφονίες εις βάρος ε, των ε, ε, δημοσιογράφων. Υπάρχει ένα διμερές θέμα με την Βρετανία που εκκρεμεί και δεν δίνεται στη συμφωνία για την έγκρισή σα. Η ε, Ρωσία έχει μεγάλο φυσικό πλούτο, αντιμετωπίζει δημογραφική βέβαια κρίση. Η οικονομία της είναι σε πολλά επίπεδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το θέμα του Ιράν, ε, τη διάδοση των όπλων για την Κορέα, για τα Βαλκάνια. Χρειαζόμαστε απαραίτητα την υποστήριξη σας. Γι' αυτό εγώ στηρίζω την ένταξη της ε, Ρωσίας στον ΠΟΕ. Βέβαια έχω κάποιες ε, αμφιβολίες για τις προξενικές θεωρήσεις, παρότι εμείς σε εμά, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, καλά θα ήταν να σας δώσουμε θεωρήσεις, να έχονται περισσότερο όσοι να ψωνίζουν στο Χάροντς. Πάντως, το να δίδονται διπλωματικά διαβατήρια στην Μολδαβία, ε, στην υπερδνηστερία, στην ε, Μολδαβία. Καλό αυτό, αλλά δεν δέχεστε όμως να πάνε οι παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία για να παρακολουθήσουν ε, καταγγελίες για εθνοκάθαρση στα κατεχόμενα εδάφη. Επίσης, άκουσα ότι η Ρωσία δεν θέλει να υπογράψει το ενεργειακό κεφάλαιο. Η Ουκρανία το έκανε αυτό προς τιμήν τη και δέχτηκε να υπάρχουν ε, και άμεσες ε, διμερείς επενδύσεις ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή λοιπόν η συγκεκριμένη κίνηση είναι ένα πολύ συγκεκριμένο δείγμα αμοιβαία εμπιστοσύνη, αν δηλαδή και η δική σα κυβέρνηση υπέγραφε το ενεργειακό κεφάλαιο και τα επιπρόσθετα κεφάλαια που θα έδιναν πρόσβαση σε ευρωπαϊκέ επενδύσει και κυρίω στον αγωγό τη Gazprom. Υπάρχουν πολλά θέματα. Λίγα εγώ σας είπα για να τα σκεφτείτε. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Ο κύριος Αγκουράκης παρακαλώ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να εκφράσω στον πρέσβη Τσιζόβ ε, τα συλληπιτήρια της ομάδας μας και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για ε, μια ερώτηση που μας απασχολεί πάρα πολύ. Επειδή έγινε πολλή συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα ήθελα να σας πω ότι με αγανάκτηση εγώ τουλάχιστον διαπίστωσα ότι το ΝΑΤΟ υιοθέτησε ένα νέο δόγμα, ένα νέο επιθετικό δόγμα το οποίο στρέφεται κατά των λαών όλου του κόσμου και σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, σε καμία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δεν πέρασε αυτό το δόγμα από, από κανένα εθνικό κοινοβούλιο. Γι' αυτά οι συζητήσει, γι' αυτό το λόγο οι συζητήσει περί ανθρώπινων δικαιωμάτων κτλ. πρέπει να είναι σε πιο χαμηλού τόνου σε αυτή την αίθουσα, διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα δημοκρατία. κατά την άποψη μου. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, δεν θέλω να επεκταθώ. Αλλά σε σχέση με το ζήτημα αυτό, ένα ζήτημα που μα απασχολεί πάρα πολύ είναι το θέμα τη ειρήνης και τη ασφάλεια. Και η ερώτησή μου στον κύριο Πρέσβη είναι πολύ συγκεκριμένη. Τι άλλαξε στην αντιπυραυλική ασπίδα του ΝΑΤΟ, ώστε να οδηγήσει τη Ρωσία σε μια διαφορετική θέση στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Θυμόμαστε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια μεγάλη αντίδραση από λαούς και εργαζόμενους αλλά και από τη Ρωσία στην Αμερικάνικη αντιπυραυλική ασπίδα. Τώρα έχουμε μια καινούρια αντιπυραυλική ασπίδα. Οι στόχοι είναι οι ίδιοι, οι απειλές είναι οι ίδιε, η Ρωσία έχει αλλάξει θέση. Αν μπορούσε ο κύριος Πρέπει να μου εξηγήσει τη θέση του. Ευχαριστώ. Grazie signor eh, onorevole Angurakis. Mm, per ehm, rispettare Ευχαριστούμε τον κύριο Αγκουράκη. Κοιτάξτε, για να κρατήσουμε το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να περιορίσω κατά το ίμιση το χρόνο παρέμβασης ε, των επόμενων ομιλητών. Ε, θα πρέπει να δώσω βέβαια και 10 λεπτά ε, στους πρέσβεις για να απαντήσουν. Υποβλήθηκαν πάρα πολλές ερωτήσεις. Κύριε Πέτρε, λυπάμαι, εσείς ένα λεπτό. Εγώ θα ήθελα ε, να εκφράσω επίσης ε, τη συμπαραστασή μου, τα συλληπιτήριά μου στα, στους συγγενείς των θυμάτων. Εμείς είμαστε μέλη της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας ε, με τη Ρωσία και ελπίζουμε κάτι τέτοιο να συνέβη τελευταία φορά. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε για μια στρατηγική συμφωνία που λέμε ότι είναι απαραίτητο να εργαστούμε σε όλα τα επίπεδα. είναι απαραίτητο να προχωρήσει ο εξυγχρονισμός. Ο πρόεδρος κ. Μετβέντεφ το είπε και μόνος του ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί η κοινωνία. Εγώ είμαι για δεύτερη φορά μέλος αυτής της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου, άρα δηλαδή έχω εμπειρία και μπορώ να πω ότι μιλάμε ανοιχτά. Μερικές φορές λέγονται και σκληρά λόγια. Δεν υπάρχουν πια θέματα ταμπού. Εντάξει, δεν είμαστε πάντα ικανοποιημένοι με ε, τις συνέπειες ε, των συζητήσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις συζητήσεις για να επιτύχουμε μεγαλύτερη συνένεση ε, στα βασικά θέματα της συμφωνίας. Η βάση της συμφωνίας είναι βέβαια οι αξίες και οι αρχές. Σήμερα ελέγχθησαν τόσα πολλά που εγώ δεν θέλω να εμβαθύνω στο θέμα αυτό. Θέλω όμως ε, να υποβάλω μια ερώτηση και στους δύο διαπραγματευτές. Εσείς την κατάσταση πώς την αξιολογείτε πόσο έχουμε προχωρήσει στο θέμα του εξυγχρονισμού, σε αυτά που πραγματικά χρήζουν εξυγχρονισμό. Γιατί από την αποτελεσματικότητα των διαπραγματεύσεων εξαρτάται και η λειτουργία της ε, συμφωνίας. Ο κύριος Γιακονσάη. Η κυρία, με συγχωρείτε. Κυρία Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, έχει υπάρξει ποιότητα, βελτίωση της ποιότητας, ε, κυρίως σε επίπεδο νέων. Σήμερα έρχονται πολλοί νέοι από τη Ρωσία ταξίδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δείξω ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό ε, για την κοινωνία των πολιτών. Ε, η αμοιβαιότητα είναι καθοριστικό στοιχείο. Οι Ρώσοι αγοράζουν ιδιοκτησία στην Ευρώπη, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τους Ευρωπαίους. Πολύ δύσκολο να αγοράσουν αυτή η ακίνητα στη Ρωσία. Οι Φινλανδοί έχουν πρόβλημα. Δεν, μπορούμε εμείς να αγοράσουμε ακίνητη περιουσία στη Ρωσία. Και γι' αυτό ερωτώ τόσο τον κύριο Σόλβαν όσο και τον Ρώσο πρέσβη. Αυτή η αμοιβαιότητα, μα δεν μπορείτε να την προάγετε περισσότερο στι διαπραγματεύσεις σας. Ευχαριστούμε την κυρία Γιακονσάρη. Ένα λεπτό, Μαντλενέρ. Θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος του Ολλανδικού Κόμματος Ελευθερίας και επιτρέψτε μου να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου ε, στα θύματα της επίθεσης ε, στο αεροδρόμιο της Μόσχας. Ε, πρέπει να σας πω ότι έχουν υπάρξει εξελίξεις. Ε, Εν τω ε, μπορώ να έρθω σε επαφή με φίλους μου στη Ρωσία που μιλάνε αγγλικά. Η Ρωσία χρειάζεται την Ευρώπη και η Ευρώπη τη Ρωσία και εγώ ε, θα ήθελα να ενθαρρύνω τους διαπραγματευτές. Κάποιες παρατηρήσεις για τους δύο πρέσβεις. Η αντιμετώπιση του μουσουλμανικού, της μουσουλμανικής τρομοκρατίας. Κοιτάξτε, οι Ολλανδοί έχουν πρόβλημα με τη διάδοση της ε, μουσουλμανικής θεωρίας που δεν είναι συμβατή με τη δημοκρατία. Και νομίζω ότι η Ευρώπη έκανε τεράστιο λάθος αναγνωρίζοντας το κοσφοπέδιο. Ε, το κόμμα μου ε, λυπάται αλλά και ανησυχεί πάρα πολύ. Η Ολλανδία ανησυχεί και για το καθεστώς στο Ιράν. Η απειλή από το Ιράν είναι όλο και μεγαλύτερη και ελπίζω η Ευρώπη και η Ρωσία από κοινού να αντιμετωπίσουν τον κύριο Αχμαντή Νικολά, Νικολάη, για ένα λεπτό. Πρέπει να αγνοήσουμε, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε μάλλον κάποια μηνύματα. Ε, διαφορετικά δεν θα ανταποκρίνονται οι διαπραγματεύσεις στην πραγματικότητα που επικρατεί. Δεν θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στα όσα υπόθηκαν στο συνέδριο των Παρισίων, αλλά θα πρέπει να να θέσω δύο ερωτήσεις. Ποια είναι η αποψή σας σχετικά με τη συνεργασία στις θέματα γεωργίας και μια άλλη ερώτηση που νομίζω πως έχει ήδη τεθεί, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία που συνεχίζει να αποτελεί μια συνολική απειλή. Ο λόγο του κ. για να Συνάδελφοι, και εγώ εκφράζω ε, τα συλληπιτήριά μου προς τους ε, ε, Να πω λοιπόν ότι επειδή έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό ε, θα περιορίσω τις ερωτήσεις μου. Απευθύνομαι προς τον κύριο Οσάλβαν σχετικά με τις ε, προξενικές θεωρήσεις. Αυτό το καθεστώς υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω το εξής. Η Κομισιόν έχει κάνει κάποια ανάλυση αυτής της ε, χρονικής περίοδου. Πετύχαμε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα από τη διευκόλυνση στις θεωρήσεις. Υπάρχει κάποια ισορροπία στους αριθμούς Ρώσων που έρχονται στην Ευρώπη και αντίστροφα. Γιατί εγώ δεν νομίζω ότι είναι ισορροπημένη αυτή η σχέση. Ε, και ποια είναι η, το κοινωνικό υπόβαθρο των επισκεπτών. Κύριλοβ, ε, και θα κλείσει έτσι ο γύρος των ερωτήσεων για ένα λεπτό. Εγώ, Πρόεδρε, αν είναι βέβαια δυνατόν, επειδή υποβλήθηκαν πάρα πολλές ερωτήσεις, εγώ θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου στις σειράξεις που έχουν προκύψει. Γειτονία. Ε, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει. Ε, θα με ενδιέφερε να γνωρίζω, να μάθω κατά πόσο μπορούμε να συνεργαστούμε για να ε, αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον μία από τις δύο ε, παγωμένες σειράξεις όπως αναφέρονται εισαγωγικά. Ας πούμε, τον Αγκόρνο Καραμπάχ είναι μια τέτοια περίπτωση ή είναι μια ε, παγιωμένη περισσότερο σύραξη που υφίσταται εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κάθε ένας από τους δύο προσκεκλημένους μας ε, έχουν 10 λεπτά, έχει 10 λεπτά στη διάθεσή του. Ε, θα λάβουν το λόγο όπως ακριβώς ξεκίνησαν ο κύριος Σάλιβαν και θα ακολουθήσει ο Ρώσος πρέσβης. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας. Υπάρχουν ένα-δύο στοιχεία για τα οποία, δύο, δύο, για τις οποίες δεν έχω ε, τα, στα έγγραφά μου σήμερα εδώ τις απαντήσεις. Θα το μελετήσω και θα σας ενημερώσω βεβαίως. Τώρα, κοιτώντα τα διάφορα θέματα που αναφέρθηκαν, και για το θέμα της ε, πρόσβασης ε, στον ΠΟΕ. Έχετε δίκιο ότι δεν είμαστε μόνοι στον ΠΟΕ και αυτή είναι η ίστατη, ο ίστατος οργανισμός συνένεσης ανάμεσα σε 153 χώρες. Οπότε οποιαδήποτε διαδικασία προσχώρησης είναι περίπλοκη και μπορούμε να προβλέψουμε ότι πολλές χώρες θα έχουν θέματα δικά τους να θέσουν και εμείς μπορούμε να ενεργήσουμε ως ε, διαμεσολαβητής, με διευκολυντής των διαπραγματεύσεων. Έχουμε επιρροή στον ΠΟΕ και είναι Πολύ όμορφη η συμμετοχή και είναι πάντως θέμα στρατηγικής σημασίας για μας και όχι μόνο ευχαρίστως θέλουμε να ολοκληρώσουμε τις διμερείς μας συμφωνίες αλλά ευχαρίστως θα συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς και άλλους για να διευκολύνουμε την ε, διαδικασία. Φυσικά η Ρωσία θα πρέπει να βρει και τις λύσεις με άλλες, τις άλλες χώρες που έχουν προβλήματα. Είναι περίπλοκη διαδικασία αλλά νομίζω πως είναι ιστορική σημασίας. Γιατί θα πρέπει να μείνουμε απαθείς σε αυτή τη διάσταση, γιατί είναι η τελευταία μεγάλη οικονομία που δεν ανήκει στο σύστημα ΠΟΕ, πράγμα το οποίο θα είναι πηγή μεγάλου ωφέλους και ευημερία για την κοινότητα του ΠΟΕ. Κυρία Σαλαφράγκα, για το θέμα των θεωρήσεων. Νομίζω πως όλοι γνωρίζουμε την λεπτότητα του θέματος και υπάρχει χωριστή διαδικασία για τη συζήτηση του θέματος αυτού, επειδή ακριβώς είναι τόσο ιδιαίτερο και θα πρέπει να δούμε πού, πού, κατευθυνόμαστε, τι πρέπει να μπει μέσα σε αυτή τη συμφωνία. Οπότε δεν έχουμε προκαθορισμένες ιδέες, δεν είναι κάτι το οποίο θα διαπραγματευτούμε σε αυτό το πλαίσιο, αλλά είναι ξεκάθαρο πως είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα για τη ρωσική πλευρά, όσο και για μας, όπως αναφέρατε πολύ, και είναι σαφές ότι από τη στιγμή που θα έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουμε αυτό να το αντικατοπτρίσουμε και στη συμφωνία και να αποφασίσουμε σε ποιο βαθμό οι αναφορές μας και οι παραπομπές μας στη συμφωνία και στο βαθμό που θα είναι πλήρη συμφωνία για τις θεωρήσεις ή αν θα είναι δύο διαφορετικές δηλώσεις προθέσεων. Για το θέμα των στατιστικών για τις θεωρήσεις και τα πολύ σημαντικά θέματα που αναφέρατε, δεν έχω σήμερα μαζί μου τις απαντήσεις, αλλά φυσικά θα Έχουμε έναν ε, ενεργό διάλογο περί όπου εξετάζουμε όλα αυτά τα θέματα και θα σας διαβεβάσουμε τις σχετικές πληροφορίες. Για το θέμα της κυρίας Όμεν Ρόιτεν, για το Τελωνιακή Ένωση, πολύ περίπλοκο θέμα. Το παρακολούθησα στενά όσο ήμουν και στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Νομίζω πως ε, με όλο το σεβασμό ε, κύριε Πρέσβη, δεν καταλαβαίνουμε όλες τις επιπτώσεις μιας τέτοιας θελωνιακής ένωσης για τις διμερείς μας σχέσεις και για την πρόσβαση στον ΠΟΕ της Ρωσίας. Το Καζακστάν και η Λευκορωσία θέλουν να έχουν τελωνιακή ένωση μαζί μας, αλλά πρέπει καλύτερα να καταλάβουμε ακριβώς τις νομικές επιπτώσεις για τις διμερείς μας ε, ρυθμίσεις, αλλά και το πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει στον ΠΟΕ και ζητήσαμε τους Ρώσους συναδέλφους να μας δώσουν λίγο περισσότερες πληροφορίες και γι' αυτό και εδώ ίσως θα πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο τις συζητήσεις μας στο κεφάλαιο εμπόριο και επενδύσεις. Για το θέμα των αξιών. Φυσικά και είναι θεμελιώδης. Αν Και φυσικά δεν μου αρέσει να διαπραγματεύομαι μέσα σε περιστάσεις όπου δεν είναι σαφής η συμφωνία για όλα αυτά. Ωστόσο έχουμε κοινέ αξίες και η ιδέα είναι όλα αυτά να επιβεκυρωθούν μέσω μιας συμφωνίας. Δεν συμφωνούμε στα πάντα, αλλά ελπίζουμε ότι έτσι θα έχουμε μια αμοιβαία συμφωνία. Βέβαια, μια τέτοια ε, διαπραγμάτευση και μια τέτοια είδου συμφωνία χρειάζεται και μια συμβιβαστική, ένα συμβιβαστικό πνεύμα. Δεν θα δεχτεί μονομερή λύση, ούτε θα δεχτούμε εμεί μείωση τη δέσμευσή μα για συγκεκριμένε αρχέ. Μπορούμε τώρα να τετραγωνίσουμε αυτόν τον κύκλο και να φτάσουμε στη συμφωνία. Πιστεύω πω ναι, αλλά θα είναι λίγο δύσκολο και πρέπει να συνεχίσουμε την εργασία μα για αυτό το θέμα. Πάντω πιστεύω είναι κοινή η δέσμευσή μα να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση. Ο πρέσβης το αναγνώρισε και ότι θα είναι ένα, μια από του τομεί όπου το Κοινοβούλιο θα επαγρυπνεί. Και εγώ ως διαπραγματευτής το γνωρίζω αυτό και γνωρίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Uh, Κύριε Σούλτς, μιλήσατε για το θέμα των διαφόρων τμήματων, ε, οργάνωση, ισχύουσα συμφωνία και ούτω καθεξής. Δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε από αυτά και μάλιστα η κυρία ήταν, ρώτησε την ίδια ερώτηση, αν θα είναι αυτό εμπόδιο. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω πως προσπαθούμε να φτιάξουμε στα να βασιστούμε σε αυτά που έχουμε, αλλά να φτιάξουμε μια πιο νέα και πιο καθολική συμφωνία. Και δεν νομίζω πως η συνεχιζόμενη συνεργασία αποτελεί εμπόδιο γι' αυτό. Συμβάλλει αντίθετα στην καλύτερη κατανόηση και σε μια κοινή αίσθηση σκοπού, στόχου, κοινών στόχων. Για το θέμα το εξυγχρονισμό δεν έχουμε συμφωνία, γι' αυτό έχουμε την εταιρική σχέση, είναι ένα σημαντικό τμήμα της σχέσης μας και θα θέλαμε να βασιστούμε σε αυτό για σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία. ώστε να συμβάλλουμε στον εξυγχρονισμό της Ρωσίας που στο κάτω-κάτω της γραφής είναι θέμα ρωσικό το πώς θα προχωρήσει και πώς θέλει να εξυγχρονιστεί και αν θέλει. Για το θέμα τώρα της συνεργασίας στη Γεωργία... Δεν έχω τις λεπτομέρειες της φύσης της συνεργασίας για τη Γεωργία και θα επανέλθω με απαντήσεις, αλλά θα υπάρχει ένα τμήμα. Και τέλος, για το θέμα των παγωσμένων γειτονικών συγκρούσεων που είναι πολύ λεπτό και σημαντικό, να σας πω ότι τελικά είναι μια συμφωνία πλαίσιο. Δεν θα δώσει τη λύση για τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, αλλά ελπίζουμε ότι θα, θα οικοδομηθεί έτσι η εμπιστοσύνη και θα αποτελέσει αυτή η συμφωνία τη βάση για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα στο μέλλον. Φυσικά, καθώς προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις, η πρόοδος σε αυτά τα μόνιμα προβλήματα θα βοηθούσε. υπάρχει ε, άμεση σύνδεση μεταξύ της λύσης αυτών των παγωμένων συγκρούσεων και της ε, ολοκλήρωσης αυτών των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, είναι στρατηγική σημασία σε αυτές οι διαπραγματεύσεις. Ε, Εμεί συνδέομαστε με τη Ρωσία με πολλές κοινέ αξίες, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, ε, γεωγραφικά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να πετύχουμε ένα ποιοτικό άλμα ε, στη σχέση μας, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που είναι υπαρκτά, που πολύ τα αναφέρατε και που αποτελούν ζήτημα ε, στα όρια των διπλωματεύσεων που περιπλέκουν ε, τις διπλωματεύσεις. Από την άλλη πλευρά, καμιά από τις αρχές δεν θέλει να εγκαταλείψει τις ε, πολύ αγαπημένες τις αρχές, ωστόσο θέλουμε να υπάρξει επιτυχία στις διπλωματεύσεις. Και τώρα, αν θα είμαστε εμεί, ή ο πρέσβης Χίσοφ που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει νέου διαπραγματευτές, εγώ ελπίζω πως θα μπορέσουμε να να, γίνει, να, να ολοκληρωθούν οι διπλωματεύσεις. Από την άλλη πλευρά είμαι και ε, πολύ μετριοπαθή, Ωστόσο, πρέπει να είναι στρατηγικό στόχο για την Ένωση, για τα κράτη-μέλη μα η ολοκλήρωση και για το Κοινοβούλιο και γι' αυτό και χρειάζεται απαραίτητη επένδυση χρόνου και προσπάθεια. Τονίζω ότι η διάσταση εμπόριο και ε, επενδύσει θεωρούμε πώ δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά, αλλά με την καλή θέληση όλων θα βρούμε τρόπους να προχωρήσουμε για να κλείσουμε και τα άλλα κεφάλαια. Δυόμιση χρόνια μόνο έχουν διαρκέσει οι την ένταξη στο ΠΟΕΤ διαπραγματεύονται εδώ και 17 χρόνια. Νομίζω πως το ρεκόρ το έχουμε σπάσει με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου. Είμαστε στον 20, στο 20ο έτος διαπραγματεύσεων. Δεν νομίζω πως θα σπάσουμε τέτοιο ρεκόρ. Όχι. Νομίζω πως θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία πολύ πιο σύντομα. Γιατί η πολιτική κατάσταση και η οικονομία μας υποχρεώνουν να ολοκληρώσουμε Επιτυχώ αυτές οι διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ κύριε Σάλιβαν. Έχετε τον λόγο. Κύριε Πρέσβη Χιζόφ. Well, thank you very much. I would like... Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω όλους τους αγορητές που εξέφρασαν τα συλληπιτήρια τους για την τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο της Μόσχας. Ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, είναι ένα βασικό στοιχείο της συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα την προαγάγουμε περαιτέρω και θα συμπεριλάβουμε το κεφάλαιο αυτό στη Νέα Συμφωνία τώρα. Για τον ε, εξυγχρονισμό θα σας πω πώς ε, βλέπουμε τη δομή Νομίζουμε ότι η μελλοντική συμφωνία θα αποτελεί τη νομική βάση. Και θα έχουμε και τον οδικό χάρτη, ο οποίος θα μας οδηγεί στην δημιουργία κοινών χώρων. Εταιρική σχέση για τον εξυγχρονισμό. Συμφώνω με τον Ντέιβιτ δεν είναι μια χωριστή συμφωνία, αλλά αυτό το οποίο έχουμε τώρα είναι το επωνομαζόμενο ένα ε, κυλιόμενο πρόγραμμα που υπάρχει, που λειτουργεί ως πρόγραμμα αλλά και ως ε, τρόπος εποπτείας των ε, εξελίξεων. Ή τώρα, μετά τη Λισαβόνα πραγματικότητα, οδήγησε τον κόσμο στο να εξετάσει καλύτερα και να αντιληφθεί καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δομές της, αλλά σε κάποιες διαφοροποίησεις θέματα οργάνωσης. Δηλαδή ποιος θα είναι ο συντονισμός για την εταιρική σχέση, τον εξυγχρονισμό από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση με το ότι ο κ. Μιγκερέλε εγκατέλειψε αυτή την θέση και ανέλαβε νέα καθήκοντα. Τώρα, εταιρική σχέση για τον εξυγχρονισμό δεν είναι κάτι που αντανακλά την ε, γνωστές ε, απόψεις ότι δηλαδή η Ευρώπη είναι ο απομηχανής που θα κατέλθει και θα εξυγχρονίσει την Ρωσία. Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στην αμοιβαιότητα, κάτι που είπαν οι αγορητέ. Χρειάζεται λοιπόν να αντιμετωπιστούν παρόμοιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η Ευρώπη και η Ρωσία δεν ε, είναι δύο οντότητες ε, από μόνες τους βρίσκονται και ζουν μέσα σε έναν κόσμο περίπλοκο και ο οποίος αλλάζει μέρα με τη μέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, για να παραμείνουμε σημαντικός, για να παραμείνει σημαντικός παίκτης η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει εταίρους και η Ρωσία προσφέρει τις δυνατότητες που έχει στον τομέα του εξυγχρονισμού να καταστήσει στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θέματα που άπτονται των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερία του τύπου κλπ. Η ρωσική νομοθεσία για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πολύ πιο φιλελεύθερη από κάποιους νόμους που πρόσφατα εφαρμο... Ε, ψηφίστηκαν και εφαρμόζονται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Τάνακ, αλλά μόλις ε, αναχώρησε. Δυστυχώς αναχώρησε ο κύριο Τάνοκ, αλλά θα ήθελα να διευκρινίσω πως ε, η Ρωσία υπέγραψε το 1994 την χάρτα για την ενέργεια, δεν επικυρώθηκε όπως και δεν επικυρώθηκε από άλλα κράτη που, όπως η Νορβηγία που είναι σημαντικός ενεργειακός παίκτης και τα πρωτόκολλα δεν υπάρχουν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και ε, η χάρτης ε, δεν ε, επικυρώθηκε, δεν τέθησε ισχύ. Από τότε, κατά την άποψή μας, η σημασία του έχει εκπνεύσει και έχει λήξει και συζητάμε με άλλους εταίρους, με τον ΟΗΕ κλπ περί μιας νέας ε, αντίληψης της ενεργειακής συνεργασίας βασιζόμενης σε αρχές που συζητήθηκαν το, στον Αγία Πετρούπολη 2006. Τώρα για τις προξενικές θεωρήσεις. Προσωπική μου άποψη νομίζω ότι στην ε, σύγχρονη Ευρώπη οι θεωρήσεις αποτελούν αναχρονισμό αντιλαμβανόμαστε πως αυτό είναι περισσότερο πολιτικής φύσης ζήτημα και λιγότερο οργανωτικής φύσης ή τεχνικής φύσης διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να καταργήσουμε τις θεωρήσεις με κάποιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, υποθέτω. Δεν θα πρέπει να ε, το ζήτημα, αλλά κάναμε σημαντική πρόοδο πέρυσι. Αποφασίσαμε να περάσουμε από μια διαρευνητική φάση σε μια επιχειρησιακή φάση. Ομού λοιπόν με την ε, Κομισιόν ε, οστικοποιούμε μια σειρά από κοινά βήματα τα οποία θα πρέπει να αντιληφθούν προκειμένου να καταργηθούν οι προξενικές θεωρήσεις ε, για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Έχω κάποια στοιχεία για πέρυσι. Ο αριθμός ήταν περίπου 4 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια Ρώσοι επισκέφτηκαν, δεν θα έλεγα, τις ε, χώρες του Σέγγιν και 1,5 εκατομμύρια πολίτες του χώρου Σέγγεν που επισκέφθηκαν τη Ρωσία. 2,5 και 1,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία μπορούν να σας κάνουν να καταλάβετε την διάσταση του ζητήματος. Ισλάμ, Ιράν, ε, δεν θα ήθελα να θίξω το Ιράν να πω ότι συνεργαζόμαστε στενά και με τις Ιρανικές αρχές και με την Κάθριν Άστον και με άλλα κράτη που ονομάζονται 3 ε, συν 3 ή 5 συν 1, αλλά με στόση 6 είναι οι συμμετέχοντες και είχαμε μια συνάντηση πριν από μερικές μέρες στην Κωνσταντινούπολη. Φυσικά δεν είχαμε και ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά δεν ε, ήταν και αποτυχία αυτή η συνάντηση. Τώρα για το Ισλάμ, ίσως να εκπλαγείτε ότι η μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα στην ε, Ευρώπη είναι η Ρωσική Ομοσπονδία. Έχει τον μεγαλύτερο αριθμό μουσουλμάνων στην Ευρώπη, άνω των 20 εκατομμυρίων και έχει μια παράδοση χιλιετίας ε, συνύπαρξης, χιλιετούς συνύπαρξης της πλειοψηφίας των ε, χριστιανών Ορθοδόξων και των μουσουλμάνων και δεκάδων άλλων ε, θρησκευτικών ομάδων. Φυσικά εδώ δεν θα ήθελα να θέσω ερωτηματικό ανάμεσα στις σχέσεις τρομοκρατίας Ισλάμ οι τρομοκράτες δεν έχουν χώρα δεν έχουν θρησκεία. Τώρα η να Καραμπάχ και η Περνιστηρία αναφέρθηκε στο πλαίσιο των θεωρήσεων. Κοιτάξτε, όταν η Σοβιετική Ένωση έπαψε να υφίσταται, υπήρχαν πολίτες της Σοβιετικής Ένωσης που παρέμειναν στα εδάφη με τα παλαιά έγγραφα ταυτότητας. Η παράταση ισχύω ε, παρετάθη για, σε κάποιες, για κάποιες περιόδους και η Ρωσική Ομοσπονδία ενέκρινε την μηδενική επιλογή. Δηλαδή, οι παλιοί πολίτες που βρίσκονται στον ε, επικράτειο της ε, Ρωσικής Ομοσπονδίας αυτομάτως ε, γίνονται Ρώσοι πολίτες. Και αυτό ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα που θα έπρεπε να γίνει. Αλλά όχι όλες οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες ακολούθησαν αυτήν την διαδικασία. Θα, θα αναφερθώ στην Λετωνία και τη Λιθουανία που επέλεξαν ε, το λεγόμενο μη πολίτες ε, της ε, Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο πληθυσμός της Απχαζίας, της Υπερνηστερίας που παρέμεινε με τα παλιά έγγραφα ταυτότητας δεν επιθυμούσαν οι περισσότεροι ή δεν τα σε οι περισσότεροι δεν επιθυμούσαν να πάρουν ταυτότητες από την Γεωργία ή την Μολδαβία. Και όταν ε, τα παλιά χαρτιά τους ε, εξέπνευσαν τότε δεν είχαν πλέον κάποιο έγγραφο επίσημο, κάποια ταυτότητα. Και θα έπρεπε να υποβάλουν έτοιμα στην Ρωσική Ομοσπονδία. Στην υπενδυστερία ορισμένη υπέβαλαν στην ε, Ουκρανία. Και σήμερα η πλειοψηφία του πληθυσμού αυτών των τριών εδαφών έχουν ρωσικά διαβατήρια. Δύο από αυτά έχουν ε, αναγνωριστεί ως ε, ανεξάρτητα κράτη και η υπερδυστερία προσβλέπει σε μια ειρηνική επίλυση του προβλήματος με τη Μολδαβία, αλλά σε ό,τι αφορά τις θεωρήσεις και τα διαβατήρια δεν μπορούμε να αγνοούμε την ε, χορήγηση ρουμανικών διαβατηρίων σε πολίτες Μολδαβίας. που μερικές φορές είναι ε, πολύ μεγαλύτερος από τον ίδιο τον πληθυσμό των, ε, της υπερνηστερίας. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, η αντιπυραυλική ασπίδα των ΗΠΑ ερώτηση του κ. Αγκουράκη. Αυτό είναι ένα χωριστό ζήτημα, θα προσπαθήσω να είμαι, προσπαθήσω να είμαι μάλλον σύντομος. Αφού ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Ομπάμα, όπως γνωρίζετε, κατάργησε το προηγούμενο σχέδιο της κυβέρνησης Μπούς για την εγκατάσταση αντιπραγματικής ε, ασπίδας στην ε, Πολωνία και την Τσεχία. Και πρότεινε ένα πρόγραμμα διαφορετικό το οποίο είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τις ΗΠΑ αλλά και με άλλα κράτη του, μέλη του ΝΑΤΟ για τη δημιουργία ενός, κοινού αντιβαλιστικού συστήματος. Δεν συμφωνήσαμε σε τίποτα περί αυτού. Ακόμα και στη Λισαβόνα τον Νοέμβριο στην ε, κοινή συνάντηση που είχε ΝΑΤΟ-Ρωσία. Συμφωνήσαμε στο να συζητήσουμε το ζήτημα. Και φυσικά ε, οποιοδήποτε σύστημα αντιβαλιστικό θα είναι στρατηγικό ή υποστρατηγικό. Σε υποστρατηγικό επίπεδο έχουμε συζητήσεις ε, ε, που διαρκούν εδώ και χρόνια. και που αφορούν την προστασία κάποιων ομάδων τήρησης, ειρνητικών ομάδων που βρίσκονται την Φίλιο. Τώρα, αν το στρατηγικό, ε, το οποίο σημαίνει μια συνολική ασπίδα, ένα συνολικό σύστημα, αυτό είναι κάτι το διαφορετικό και πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Η νέα Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία START μόλις κυρώθηκε από την Βουλή της Ρωσίας και ε, έχουμε δηλώσει ότι θα εποπτεύουμε, θα ελέγχουμε ε, την τήρησή της, ε, της συμφωνίας και θα κάνουμε το συγχειρισμό με το αντιπαλιστικό σύστημα. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι ξεπέρασα σημαντικά τον χρόνο που είχα στη διάθεση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ε, και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Τσίζοφ και ευχαριστούμε βέβαια και τον δικό μας το διαπραγματευτή, τον κύριο Σάλιβαν. Ευχαριστώ όλους σας. Ε, καταλαβαίνετε βέβαια πόσο σημαντική είναι αυτή η συμφωνία Κατά τον 19ο αιώνα είδαμε ότι υπήρχαν εσωτερικές διαμάχες στην Ευρώπη και αυτές οδήγησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στον 21ο αιώνα βλέπουμε ότι διευρύνεται η συνεργασία και πέρα από τα παραδοσιακά σύνορα της Ευρώπης ε, διευρύνεται η συνεργασία με χώρες πολύ σημαντικές. Η συνεργασία πλέον πάει προς Ανατολάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι βεβαίως, όπως φαντάζομαι και εσείς όλοι, ότι οι αυτές θα και σύντομα θα έχουμε αίσιο τέλος. Η συνεδρίασή μας συνεχίζει το απόγευμα στις 3 με ψηφοφορία ξεκινάει. Θα σας παρακαλούσα να έρθετε στην ώρα σας γιατί και πάλι το απόγευμα η μερίσια διάταξη είναι πολύ επιβαρημένη και είναι πολύ σημαντικές οι συνέπειες αυτής της ψηφοφορίας. Παρακαλώ λοιπόν να είστε εδώ ακριβώς στις 3.